dear colleagues, I think we should start. Συνάδελφοι, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά από τη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην πρώτη μας ε, συνεδρίαση για φέτος, οπότε καταρχήν ακριβώς επί την πρώτη συνεδρίαση θα ήθελα να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. και ελπίζω όλα όσα επιθυμείτε να τα πετύχετε μέσα στο 2019. Περνάμε λοιπόν απευθεία στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη έτσι όπω αυτή είναι δεδομένη στο σχέδιο. Εάν όχι, αν δεν υπάρχουν δηλαδή διαφωνίε, ε, θεωρούμε πω εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνάμε στο δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών των ε, συνεδριάσεων της Επιτροπής μας από την 8η και την 15η Νοεμβρίου. Τα εν λόγω πρακτικά τα έχετε λάβει εντό του φακέλου σα για τη σημερινή συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω να ζητά κανεί το λόγο. Οπότε σα προτείνω να θεωρήσουμε ω εγκεκριμένα αυτά τα πρακτικά εφόσον δεν εκφραστούν αντιρρήσει ε, κατά τη διάρκεια της σημερινής ε, συνεδρίασης. Ε, τώρα, περνάω στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Να σας πω καταρχήν πως ε, διερμηνία σήμερα έχουμε κατά τις εξής γλώσσες. Ε, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσέχικα, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβένικα, βουλγαρικά και ρουμανικά. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ως ε, συνήθως ότι έχουμε web streaming για τη σημερινή συνεδρίαση. Επίσης να σας ενημερώσω ότι έχουμε μία νέα συνεργάτηδα στην γραμματεία της Επιτροπής Κάλτ, η κυρία Ντενίς Βαλμέρκα η οποία αντικαθιστά την ε, κυρία Βαντμούρκε, η οποία για τους λόγους της ε, περιτροπής ανάληψης καθηκόντων στην γραμματεία άλλαξε θέση. Οπότε καλωσορίζουμε θερμά τη νέα συνάδελφο στη γραμματεία και ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία της. Ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν. Μία ακόμα ανακοίνωση από τη δική μου πλευρά είναι εξή. Ε, ανάμεσα στις 10 και στις 11 ίσως να χρειαστεί να εγκαταλείψω την αίθουσα για λίγο. Ε, μην εκπλαγείτε, έχω μια διμερή συνάντηση, ε, δεν θα αργήσω, η κυρία Βόσκοβα θα με αντικαταστήσει ε, για όση ώρα λείψω και μην ανησυχείτε, ε, θα είμαι ε, στην ώρα μου εδώ για να περάσουμε στη συζήτηση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Ας περάσουμε τώρα στις προτάσει ε, που έχουμε για τι ειδικέ ψηφοφορίε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη από αυτέ, την απαλλαγή 2017, Γενικό ε, Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Τρογεύσκη ήταν ο για αυτή την γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια προκατακτικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ όλου του συνάδελφου ε, θερμά Και βλέπετε ότι έχουν υποβληθεί πολύ λίγε τροπολογίε. Ε, αυτό καταδεικνύει την πολύ καλή συνεργασία που κάναμε και ευχαριστώ πραγματικά όλου ε, του ε, συναδέλφου και του κοιόδη συζητητέ για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε που μα επέτρεψε να καταλήξουμε γρήγορα σε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω πω το έγγραφο που έχουμε μπροστά μα σήμερα είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ θερμά, λέει Πρόεδρος, τον εισηγητή, αλλά φυσικά και τους εισηγητές και την ε, Γραμματεία και όλους τους συναδέλφους και περνάμε με την... ξεκινάμε μάλλον με την τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Όλα λαμβάνει με προφορική τροπολογία 1 σε σχέση με την τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, ε, δεν ήταν σαφές το αποτελέσμα, οπότε ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 10 ψήφους υπέρ και 8 κατά. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα γιατί καταπίπτει, οπότε περνάμε στη 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου της χρονομοδότησης ονομαστή ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Geschlossen πέρα τη ψηφοφορία. εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και καμία αποχή. Με συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία εγκρίνεται η σημερινή γνωμοδότηση και ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν σε σχέση με αυτήν. Ε, περνάμε τώρα στην ε, ε, ψηφοφορία σε ό,τι αφορά την έγκριση τη γνωμοδότηση, σε ό,τι αφορά το μεταφραστικό κέντρο των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο πάντοτε τη απαλλαγή του 2017. Και σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ε, αρμόδιο συστήκτης ήταν ο κύριος Τρογεύσκη. Δεν βλέπω όμω να ζητάει το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε απευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε και σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση στην ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου της γνωμοδότησης, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και αυτή η γνωμοδότηση εγκρίνεται με συντηρητική πλειοψηφία 18 ψήφων υπέρ και μία ψήφου κατά. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία σε ό,τι αφορά την έγκριση μια γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ενό μηχανισμού γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Ε, η κυρία Μαρία Τερέζα Χιμένε ε, Μπαρμπά, την αρμόδια ε, θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός στις σχέσεις γειτονίας. Θα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπόλοιπους ε, εισηγητές που εργάστηκαν ε, σε ένα σχέδιο που νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την ε, εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές και ξεκινούμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 και 11 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται 92 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 98 μαζί με τη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε την 105 οπότε άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 10 ψήφους υπέρ και 10 ψήφους κατά. 106 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 111 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά.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 αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 και 9 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ε, σηκώστε τα χέρια όμως να σας βλέπω. 57 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παίρναμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. 17 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τόσο εύκολη την σημερινή ψηφοφορία, γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Να το αναγνωρίσουμε λοιπόν. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της σημερινής διάταξης. Ελπίζω να έχουν έρθει η προσκεκλημένη μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε λοιπόν στο σημείο 7 της σημερισίας διάταξης. Πρόκειται για μία μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτισμού και ανέθεσε στο θεματικό τμήμα χρηματοδότηση του κινηματογράφου και ψηφιακή ενιαία αγορά. Το μέλλον, ο ρόλος της αρχής της εδαφικότητας και τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν θερμότατα τον καθηγητή Μπέρντ Χούγκενχολτς από το Ινστιτούτο Πληροφοριακού Δικαίου του Άμστερνταμ. Καλώς ήλθατε. Ο κύριος καθηγητής θα μας παρουσιάσει τα σημαντικότερα σημεία της μελέτης αυτής ε, που εστιάζει στον ρόλο της ε, εδαφικότητας ε, και τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης των κινηματογράφων. Η μελέτη αυτή μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα μοντέλα χρηματοδότησης στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χρηματοδότηση του κινηματογράφου μετά από την ψηφιακή αλλαγή καθώς και τις τάσεις ε, στη συμπεριφορά των καταναλωτών σε αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές μεθόδους χρηματοδότησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας δίνω το λόγο για περίπου 15 λεπτά έτσι ώστε να μας παρουσιάσετε την μελέτη. Κατόπιν θα περάσουμε σε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την εισαγωγή. Είναι μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω τη μελέτη αυτή για την ε, χρηματοδότηση του ματογράφου στην νέα ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω και τους ε, τρεις συνεργάτες μου, τον κύριο Γιώστ Πόρτ, ο οποίος ηγήθηκε του project αυτού, ο κύριος Χέσφον Τίλ και ο Πέτερ Λίντχαουτ. Μαζί λοιπόν ε, κάναμε την μελέτη και θα μιλήσω εξ ονόματος όλων των συνεργατών μου. Το θέμα της μελέτης είναι και το θέμα της παρουσίασης. Ελπίζω λοιπόν να βρείτε το χρόνο να διαβάσετε την ε, μελέτη ή έστω την συνοπτική της παρουσίαση. Θα περάσω λοιπόν αμέσως στα κύρια ερωτήματα που μας ζητήθηκε να εξετάσουμε. Η μελέτη λοιπόν αυτή εστιάζει στη χρηματοδότηση του κινηματογράφου και από την κέφαλη αγορά και από τις κυβερνήσεις, από το κράτος. Τα κυριότερα ζητήματα που έπρεπε να εξετάσουμε είναι ο ρόλος της εδαφικότητας, τα εδαφικά δικαιώματα της χρηματοδότησης κινηματογράφου και πώς επηρεάζεται η χρηματοδότηση από τις ε, προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Φυσικά υπάρχει κάποια ένταση ανάμεσα στην χορήγηση εδαφικών δικαιωμάτων και στην εσωτερική αγορά. Κοιτάξαμε λοιπόν τις κυριότερες προκλήσεις οικονομικού χαρακτήρα και πολιτικού. το πεδίο εφαρμογή τη ε, εδαφικότητα θα μειωθεί, θα συρρυκνωθεί μάλλον ακόμα περισσότερο από το ενωσιακό δίκαιο. Όμω η χρηματοδότηση του κινηματογράφου είναι ε, μια πολύ σημαντική πτύχη. Κοιτάξαμε λοιπόν τις εξελίξεις, τις θετάσεις και ψάχνουμε εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να πάρουν τη μορφή πολιτικής. Περνάμε λοιπόν ευθύ αμέσω στο πρώτο ουσιαστικό κεφάλαιο της ε, μελέτη. δηλαδή μια γενικότερη ανάλυση της αγοράς και των προβλημάτων που υπάρχουν, που εξηγεί γιατί η κινηματογραφική παραγωγή εξαρτάται τόσο πολύ από εξωτερική χρηματοδότηση. Έχουμε εντοπίσει δύο παράγοντες που επηρεάζουν την χρηματοδότηση. Πρώτον, οι ιδιαίτερα είναι κάτι επενδύσεις εκ των προτέρων που κάνουν την παραγωγή μιας ταινία πάρα πολύ ε, ακριβή και έπειτα η ζήτηση είναι, κάτι ε, το απρόβλεπτο. Ο παραγωγός δεν μπορεί να προβλέψει την απήχηση μιας ταινία. και εδώ λοιπόν ε, υπάρχουν προβλήματα στην χρηματοδότηση. το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης προέρχεται από, ε, προ, ε, από συμφωνίες εκ των προτέρων, προχρηματοδότησης και συμφωνίες που έχουν γίνει με διανομής ή με ε, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που αγοράζουν τα δικαιώματα προβολής της ε, Η χρηματοδότηση λοιπόν εν μέρη προέρχεται από αυτές τις συμφωνίες. Βλέπουμε βέβαια ότι οι ευρωπαϊκές ταινίε είναι κατά μέσο όρο πολύ λιγότερο επιτυχημένα σε σχέση με τις ε, αμερικανικές παραγωγές, όμως τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τρομακτικά για την Ευρώπη. Στο 2017 είχαν γυριστεί δύο φορές περισσότερες ε, κινηματογραφικές ε, ταινίες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Αμερικανικές, όμως τα έσοδα ήταν αντιστρόφως ανάλογα. Και αυτές οι τάσεις είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ. Πολλές ευρωπαϊκές ταινίες λοιπόν έχουν προβλήματα, δεν έχουν τις οικονομίες κλίμακας που έχουν οι αμερικανικές παραγωγές και επίσης δεν υπάρχει προπολογισμό για την προώθηση μιας ε, ταινία όπως οι μεγάλες ε, παραγωγέ. Οι ευρωπαϊκές λοιπόν ταινίε εξαρτώνται κατά πολύ από τις ε, καλές κριτικές. Και σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές ταινίε δεν θα μπορούσαν να είχαν γυριστεί χωρίς δημόσια χρηματοδότηση. Και στην μελέτη λοιπόν περιγράφονται οι πολιτικές στήριξης ε, της σηματογραφικής παραγωγής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επιμέρους κράτη-μέλη. Έχουμε επιλέξει 12 κράτη-μέλη, τα οποία εξετάσαμε λεπτομερέστερα. Κοιτάξαμε λοιπόν την πολιτική στήριξη του κινηματογράφου και είδαμε ότι το 2014 πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν ε, προς ε, τη στήριξη της ε, κινηματογραφικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω επιχορηγήσεων, μέσω ευνοϊκών δανείων και ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, περίπου 5% των δανείων αυτών έχουν αποπληρωθεί. Υπάρχουν όμως διάφοροι μηχανισμοί στήριξης της κινηματογραφικής παραγωγής, για παράδειγμα φοροαπαλλαγές, τα οποία χρησιμοποιούν οι ιδιωτικοί επενδυτές. Και επίσης, πολλές φορές, οι εταιρείε πολυμέσων αναγκάζονται εντό εισαγωγικών να επενδύσουν σε μια κινηματογραφική παραγωγή. Περνάμε τώρα στο κεφάλαιο 4 της μελέτης, το οποίο εστιάζει στις νομικές προκλήσεις. η παραγωγοί παραδοσιακά στηρίζονται, για, στηρίζονται στην, αποκλειστική, στην χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων διανομής για τους κινηματογράφους για να βρουν χρηματοδότηση. Και αυτό σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτό δημιουργεί εντάσεις στην εσωτερική αγορά η οποία φυσικά είναι αντίθετη στα εσωτερικά σύνορα. Αυτές βέβαια οι επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια από ε, την εφαρμογή ενωσιακού δικαίου και την άρση των φραγμών στην ε, νέα αγορά. Ε, θα θυμάστε ίσως την οδηγία για τις δορυφορικές επικοινωνίες, την οδηγία για τη φορητότητα που εγκρίθηκε πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα την πρόταση κανονισμού για, την διαδικτυα... για τις διαδικτυακές μεταδόσεις που απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την εδαφικότητα και ε, δίνει έμφαση στη χώρα προέλευσης. Επιπροσθέτως, το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί όρια στην, ε, στη χορήγηση επιδοτήσεων και είναι ακόμα μια πρόκληση που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Το δίκαιο του ανταγωνισμού, για παράδειγμα, απαγορεύει ρήτρε οι οποίε περιορίζουν τι ε, λεγόμενε παθητικέ πωλήσει σε εδάφη για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια προβολή και διανομή. Επίσης, βλέπουμε ότι η εδαφική αποκλειστικότητα είναι όλο και ε, πιο ευάλωτη στην νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει ένα πρόβλημα. Και στο κεφάλαιο 5 της μελέτης βλέπουμε ότι έχουν προκύψει αρκετές προκλήσεις εντός της αγοράς που εμποδίζουν την χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών. Η πρώτη είναι πολύ γνωστή, το διαδίκτυο είχε μεγάλη επίδραση στην χάραξη στρατηγικής και πολλά κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια το πώς θα προβληθεί και θα προωθηθεί μια ταινία μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο βέβαια έχει αυξήσει και ε, το κοινό μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Όμως αποτελεί πρόβλημα διότι μια χώρα από μόνη της δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μια τέτοια προβολή. Έπειτα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Οι λεγόμενε κουλτουριάρικες ταινίε έχουν πρόβλημα, δεν βρίσκουν αρκετή απήχηση στους νέους. Επίσης, έχει αναδυθεί μια διεθνική κουλτούρα λόγω της μετανάστευσης, λόγω της επικοινωνίας, γι' αυτό και είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που αυτό δημιουργεί στον πολιτισμό των επιμέρους τα γούστα λοιπόν δεν έχουν σύνορα. Αλλά παρά τις εξελίξεις αυτές βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών εξακολουθεί να στηρίζεται σε αυτές τις παραδοσιακές μεθόδους. Έχουν βέβαια εμφανιστεί και νέες μέθοδοι όπως το crowdfunding, όμως ε, δεν είναι αρκετά διαδεδομένες έτσι ώστε να αποτελούν ε, ουσιαστική και εφικτή εναλλακτική λύση χρηματοδότησης. Κεφαλαίο 6 και φτάνω κοντά στο τέλος ε, της ε, παρουσίασής μου. Εδώ συνοψίζεται η θέση των ενδιαφερομένων μέρων ε, και ιδίως σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς, τους διανομής, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Αυτό το πράττουμε εξετάζοντας έγγραφα θέσεων και σχόλια που έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το χάρη. Βλέπουμε σε ένα μεγάλο βαθμό συνένεσης και ίσως αυτό μην σας εκπλήσει ότι η εδαφικότητα παραμένει ουσιαστική για τις συμφωνίες προπόλησης ε, και βλέπουμε μια επιμονή στην ελευθερία της σύμβασης ε, και ένα φόβο απομάκρυνσης ε, από την εδαφικότητα. Αυτό που ακούμε ή διαβάζουμε πολύ είναι ότι η εδαφική αποκλειστικότητα είναι βασική για την πολιτιστική διαφορετικότητα στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Αυτό μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Εμεί. θεωρούμε ότι ως αντιπιχείρημα ε, μπορούμε να πούμε ότι τελικά ζημιώνει την ε, διεθνική και πανευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, εμποδίζοντα την πρόσβαση ευρωπαϊκών ε, Ευρωπαίων ακροατών και θεατών στις ίδιες ταινίες. Και τέλος περνάμε στις συστάσεις έχουμε έναν αριθμό πέντε συστάσεων. Καταρχήν αναφερόμαστε στην εδαφική αποκλειστικότητα, αν θεωρήσουμε ότι μένει απαραίτητη για κάποιο καιρό. Συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου, για τον ανταγωνισμό, μπορεί να δημιουργήσει συγκεκριμένους κανόνες ανταγωνισμού, ε, με τη μορφή των ε, εξαιρέσεων σε μπλοκ. Και έτσι μπορούμε να επιτρέψουμε να επιβιώσουν οι ρήτρες εδαφικότητας. Ε, μια άλλη εναλλακτική που πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο ελκυστική και βιώσιμη και δεν θα απαιτούσε καμία νομοθετική παρέμβαση Απλώς ε, αλλάζει η πρακτική και μετακινούμαστε από την εδαφική αποκλειστικότητα προς ε, την γλωσσική αποκλειστικότητα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι τα δικαιώματα προπόλησης αφορούν τις γλωσσικές αγορές ε, παρά τις εδαφικές αγορές. Και το καλό της Ευρώπης ε, είναι ότι έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό γλωσσών ε, όσο και αριθμό κρατών μελών. Και αυτό θα έδινε μια καλύτερη και πιο ευρωστηνομική εναλλακτική, η οποία ε, ουσιαστικά δεν θα θυγόταν από τον δίκαιο του ανταγωνισμού και τις ανησυχίες για τις εσωτερικές αγοράς, αλλά βέβαια θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κάποιες πρακτικές και θα χρειάζονταν κάποιες αλλαγές. Επίσης, τα συστήματα στήριξης θα πρέπει να απευθύνονται περισσότερο ε, σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες και διεθνικούς πολιτισμούς. Επίσης, ε, να ξανασκεφτούμε ε, την νομοθεσία σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση από φορείς, ραδιοτηλεόραση στην εθνική νομοθεσία και επίσης ε, προτείνουμε οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στήριξης να είναι πιο επιλεκτικέ, ε, δηλαδή να υπάρχει υψηλότερος προπολογισμό για λιγότερε ταινίε ε, και για τη διανομή και την πρόθεσή τους. Αυτά έχουμε να πούμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσίαση της μελέτης η οποία νομίζω πως μας δίνει μία σειρά από ερεθίσματα για σκέψη ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του κινηματογράφου καθώς η αίσθηση που αποκομίζουμε είναι ότι πραγματικά δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για ταινίε κινηματογραφικέ. Πραγματικά με εξέπληξε αυτό ο αριθμό των 4,20 ευρώ ανά κάτοικο. Ε, ενώ ταυτόχρονα όμω δεν καταλήγουν όλε αυτέ οι ε, ε, οι ταινίες στους πολίτες μας. Οπότε θα πρέπει να αναλογιστούμε λίγο τι σημαίνει αυτό ακριβώς για μας. Περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων και βλέπω ήδη εδώ τους πρώτους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Helga Triple είναι η πρώτη. Παρακαλώ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την μελέτη αλλά και για τα πορίσματα και τις συστάσεις της. Θα ήθελα να ξεκινήσω με, κάποιες, ε, με κάποια σχόλια και μετά να περάσω σε ερωτήματα. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε την εκπόνηση αυτής της μελέτης ήταν αυτοί οι αντιφατικοί στόχοι που υπάρχουν. Δηλαδή από τη μία πλευρά να έχουμε καλύτερε ευρωπαϊκέ ταινίε και από την άλλη πλευρά με την ψηφιακή επανάσταση να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση σε αυτέ την Ευρώπη. και το πώ βέβαια μπορούμε να το επιτύχουμε γιατί γνωρίζουμε πω οι Αμερικανοί έχουν ε, τα απαραίτητα χρήματα για να λαμβάνουν ε, τι άδειε αυτέ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τι ταινίε τους ε, σε αντίθεση με του ευρωπαίου παραγωγού. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά μου. Ε, δηλαδή αυτό που βρίσκεται σε ό,τι αφορά την εδαφική αποκλειστικότητα, το geo-blocking, το ό,τι καθεξής. Αυτό που είπατε εσείς είναι ότι αυτό μπορεί να ισχύει ή όχι αυτή η εδαφική αποκλειστικότητα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δηλαδή να δώσουμε μία απάντηση. Εσείς ως επιστήμονας δηλαδή μπορείτε να λέτε πως αυτό ισχύει ή όχι, αλλά εμείς από την πλευρά μας ως πολιτικοί θα πρέπει τελικά να βρούμε να καταλήξουμε σε μια πορεία προς τα μπροστά για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ε, και μετά να δώσω και ένα παράδειγμα. Η πολωνική ταινία Ψυχρό σε πόλεμο. Δεν είναι μια αμερικανική ταινία, είναι μια ευρωπαϊκή ταινία η οποία αναφέρεται στο σταλινισμό, στη Δύση και αφηγείται μια ευρωπαϊκή ιστορία. Και διασυνοριακά βέβαια. Και αυτή η ταινία βασίστηκε ακριβώς στο εδαφικό σύστημα καθώς δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα αυτή τη στιγμή και το crowdfunding ε, αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί και ποτέ δεν θα είναι επαρκή, σε αυτή η χρηματοδότηση γιατί δεν είναι βιώσιμο ένα τέτοιο μοντέλο χρηματοδότησης ε, γιατί δεν μπορεί να βασιστεί πάνω του κανείς ως νέος δηλαδή. Οπότε δεν είμαι πεπισμένη, λαμβάνοντα υπόψη μα και όλου του ακτιβιστέ και όλη την πειρατεία ε, ότι ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργήσει, ένα τέτοιο μοντέλο θα λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα εναλλακτικό μοντέλο προς το αμερικανικό, γιατί το αμερικανικό είναι πολύ διαφορετικό από το ευρωπαϊκό και ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για πολλά ακόμα χρόνια στο μέλλον θα υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν οράματα διαφορετικά και έχουν γίνει και αναφορές από παλιά στις Ηνωμένε Πολιτείες της ε, ε, Ευρώπης αλλά εγώ πιστεύω ότι για πολλά χρόνια και στο μέλλον θα υπάρχουν ως διαφορετικά κράτη τα οποία θα συνεπάρχουν ε, μεταξύ τους. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα μας επιτρέπει να παράγουμε καλές, καλής ποιότητας ταινίες και ένα μοντέλο για να τις χρηματοδοτούμε. και παρότι υπάρχουν ε, μία σειρά από ε, φόροι τους οποίους επιβάλλουμε, περιβαλλοντικοί φόροι και άλλου είδους ε, φόροι, πάντοτε υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά τους απαραίτητους πόρους, τα απαραίτητα κονδύλια για τον πολιτισμικό τομέα. Και κάτι που, ακόμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ποιες ακριβώς είναι οι συστάσεις σας. Γιατί αυτό που αναφέρεται εδώ είναι ε, λιγότερε ταινίε αλλά υψηλότερη χρηματοδότηση. Αυτή είναι μια σαφή σύσταση, αλλά σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα, ε, δυστυχώ δεν βλέπω να υπάρχουν ξεκάθαρε συστάσει στην έκθεσή σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong εντό εισαγωγικών, δηλαδή να δώσουμε απευθεία το λόγο στον κύριο Μπούχαν για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα τη κυρία Τρούπελ και μετά να δώσουμε το λόγο στου υπολείπου συναδέλφου. Καλώ, αυτό θα κάνουμε. Έχετε λοιπόν το λόγο. Λοιπόν, θα δώσω το μικρόφωνο σε έναν και από τους συνεργάτες μου που θα έπρεπε να είναι εδώ στο βήμα, στον ε, κύριο Γιώργο Πόρτ, ο οποίος είναι ένας από τους κύριους ε, συγγραφείς της μελέτης και επικεφαλής οικονομολόγος, καθώς η ερώτησή σας αφορά οικονομικά ζητήματα, ίσως θα ήθελα να πει δύο λόγια. Σας ευχαριστώ. Η ερώτηση για το πόσο ταινίε θα θέλαμε στην Ευρώπη είναι πολιτική, πολιτιστική ερώτηση. Δεν μπορούμε να την απαντήσουμε στη μελέτη. Εδώ εντοπίζουμε ότι υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές ταινίες ε, να φτάσουν ε, στο κοινό. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές ε, ταινίες εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το να κερδίσουν φήμη σε φεστιβάλ και από δίκτυα ε, καλλιτεχνικών κινηματογράφων. Ε, έτσι λοιπόν, ε, πολλές ευρωπαϊκέ ταινίες έχουν μόνο δύο-τρεις εβδομάδες καιρό για να κερδίσουν φήμη στους κινηματογράφους και ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέχρι θανάτου θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, αυτό το ακούμε συνεχώς. Κανένας παραγωγός βέβαια δεν θέλει να μην κάνει ταινίες, αλλά κάθε παραγωγός λέει ότι γίνονται υπερβολικά πολλές ταινίε. Ε, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε υψηλότερο προπολογισμό για λιγότερες ταινίε ε, για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην ε, ευρύτερη αγορά και να έχουμε και προπολογισμό για την πρόθεση και όχι μόνο για την παραγωγή. Αν δείτε τα νούμερα, ο προπολογισμό πρόθεση για τι ευρωπαϊκέ ταινίε είναι πολύ μικρότερο από ότι για τι αμερικανικέ ταινίε. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα λοιπόν που προσπαθούμε να περάσουμε. Όμω τώρα η ερώτηση για το πόσε ταινίε πρέπει να γίνονται είναι πολιτική ερώτηση. Παρατηρούμε πάντω κάτι ιδιαίτερα περίεργο ότι ο αριθμός ταινιών που παράγονται κατά κεφαλή στις ευρωπαϊκές χώρες είναι σε σχέση με τις μικρότερες χώρες. Δηλαδή, μικρότερες χώρες ε, ουσιαστικά δημιουργούν μεγαλύτερο αριθμό ταινιών και αυτό είναι έναντι της οικονομίας κλίμακας, ε, των οικονομικών δυνάμεων και της οικονομίας αγοράς και οξύνει το πρόβλημα. Okay. Möchten Θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω, παρακαλώ. Να έχουμε πολύ συγκεκριμένες συστάσεις ε, για το κύριο ερώτημα τη έρευνα που είναι η αδαφικότητα και ο ρόλο τη αδαφικότητας στην προπόληση. Αυτό είναι το σημείο φετήρια τη όλη έκθεση που μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε. Αυτό που βλέπουμε και νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό εδώ ότι μπορεί όλοι να ευχόμαστε ότι θέλουμε να επιβιώσει η εδαφικότητα, αλλά ταυτόχρονα μετακινούμαστε προ μια Ευρώπη που καταργεί την εδαφικότητα και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει, μα αρέσει ή όχι, είναι η δύναμη της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να κάνουμε κάποιους συμβασμούς εδώ. Μια συγκεκριμένη πρόταση που υποβάλλουμε είναι είναι να μετακινηθούμε από την κινητικότητα ε, στην αποκλειστικότητα τη γλωσσική και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά εύκολα. Και είναι και μια εύρωστη νομική λύση για ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Το σημείωσα. Τώρα το λόγο έχει η Σίλβια Κώστα για τρία λεπτά το πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνά σας εξετάσατε στο πρώτο μέρος και τις καινοτομίες ε, σε ό,τι αφορά και το κανονιστικό σκέλος ε, από τη δεκαετία του 90 και μετά στην Ευρώπη για να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια σύνθεση μεταξύ της απέτησης μεγαλύτερης ε, κυκλοφορίας και της βελτίωσης των οικονομικών συνθήκων και της ανταγωνιστικότητας. Βέβαια, εδώ θέλουμε να ενθαρρύνουμε και ε, την παραγωγική πολυφωνία και την γλωσσική πολυμορφία και να μην έχουμε μόνο ένα είδος ε, πολιτιστικής ε, απεικιοκρατίας από άλλες υπήρους που έχουν μεγαλύτερη δύναμη στη διανομή. Είδα την ανάλυση σας και Όντως ισχύει ότι υπάρχει υπερβολική παραγωγή προϊόντων που δεν ε, φτάνουν σε κρίσιμη μάζα θεατών στην αγορά. και στο νέο πρόγραμμα Media Δημιουργική Ευρώπη εμείς θέλουμε να δώσουμε περισσότερη στήριξη στην συμπαραγωγή, στην πρόθεση και θέλουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε άλλες διεθνείς αγορές πέρα από την ευρωπαϊκή αγορά. Όμως ε, μπορούμε να έχουμε και ε, ένα υπόθεμα για τον υποτιτλισμό και μπορεί να είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε ε, το δίλημα ε, που αφορά το γλωσσική αποκλειστικότητα και την κυκλοφορία στην Ευρώπη. Με ενδιαφέρει το θέμα της γλωσσικής αποκλειστικότητας, το οποίο αναφερθήκατε, γιατί έχουμε διαφορετικές γλωσσικές αγορές ως δύναμη και ως διανομή. Θέλουμε λοιπόν να, να επεκταθείτε σε αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες του Video On Demand. Ε, αναφερθήκατε στον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες και είπατε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δεύτερον, όταν εσείς λέτε συμβατική ελευθερία, δηλαδή να αφήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία, αν και γνωρίζουμε το πρόβλημα ε, που έχει το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο της ε, δαφικής αποκλειστικότητας, γνωρίζοντας ε, όμως ότι μεταμορφώνεται αυτό το μοντέλο και μπορούν να υπάρχουν μεγαλύτερα περισσότερα μέσα διανομής, δηλαδή να αφήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους ε, διανομής κτλ. Αλλά εμείς ως νομοθέτες πρέπει να εργαστούμε και επί των κανόνων για να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η συμβατική ελευθερία. Σήμερα ε, έχουμε νόμους για το copyright και συνδέονται ακριβώς στο πώς θα δημιουργηθούν ε, οι συνθήκες έτσι ώστε οι μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες να πρέπει να σέβονται τη συμβατική ελευθερία μέσα σε ένα κανόνα που να λέει ότι υποχρεούνται να προβαίνουν σε αυτές τις συμφωνίες με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να μπορούν να επενδύουν και στις εδαφικές παραγωγές. Έτσι λοιπόν ε, το ε, θέμα αυτό συνδέεται με τις συμβατικές ελευθερίες διαφορετικά δεν λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο γιατί δεν υπάρχουν τα αρχικά κονδύλια αλλά θα δημιουργούνται και μία ολική εξάρτηση χωρίς ε, κανόνες αυτών που πληροφέρουν τις πλατφόρμες αλλά δεν σέβονται την αναγνώριση. Δεν έχετε λοιπόν προσεγγίσει παρκώ το θέμα αυτό στη μελέτη σα και είναι σημαντικό θέμα. Κύριε Στρογεύσκη, α όχι, όχι, με συγχωρείτε. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο καθηγητή για την απάντηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας και το βλέπουμε αυτό και όταν μιλάμε με διανομής και παραγωγούς ε, ότι χρειάζεται να βρεθεί μια ευέλικτη λύση σχετικά με ε, το ελεύθερο περιεχόμενο. Το κατανοούμε λοιπόν αυτό. Ταυτόχρονα όμως, και νομίζω πως αυτό είναι το κυριότερο μήνυμα ή έστω ένα από τα κυριότερα μήνυματα της μελέτης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενωσιακό δίκαιο. Δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτό και να πούμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή ότι δεν δεχόμαστε την εδαφικότητα σε ε, άλλους τομείς του εμπορίου εκτός ε, από αυτόν. Τώρα εντάξει υπερβάλλω κάπως, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε αυτό το γεγονός. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η εδαφικότητα αργά ή γρήγορα θα πρέπει να υποκύψει ε, στις απαιτήσει της ενιαίας αγοράς, η γρηγορα θα πρεπει να υποκυψει στις απαιτησεις της ενιαιας αγορας η οποια δεν αναγνωρίζει σύνορα. Και γι' αυτό στη μελέτη παρουσιάζουμε μία σειρά εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ε, κινηματογραφικής βιομηχανίας, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσει της ε, ενιαίας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Στρογεύσκη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας κάνω τις ερωτήσεις μου στα πολωνικά λοιπόν. Πρώτον, υπάρχει ένας μύθος στην Ευρώπη που πρέπει να διαψεύσουμε ότι η κινηματογραφική παραγωγή στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι προσανατολισμένη στο κέρδος, δεν είναι ποιοτική και ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις. Όμως αυτό δεν ισχύει. Η πολιτεία της Καλιφόρνια για παράδειγμα, χορηγεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε κινηματογραφικές παραγωγές. Ε, δεν ισχύει λοιπόν ότι οι εμπορικές παραγωγές στις Ηνωμένε Πολιτείες ανταγωνίζονται την ε, παραγωγή στην Ευρώπη. Έπειτα, δεν υπάρχει η θέληση για να χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκές παραγωγές έτσι ώστε να προωθηθούν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η αναλογία είναι, της χρηματοδότησης είναι 10 προ 1. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν εξοδεύουν 10 φορέ περισσότερα χρήματα από του Ευρωπαίου Παραγωγού για να προωθήσουν τι ταινίε του. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Πρώτον, Έχετε εξετάσει τις ε, περιπτώσεις παράνομης ε, χρηματοδότησης κινηματογραφικών ε, παραγωγών στην Ευρώπη. Ορισμένες φορές δεν απορροφώνται κονδύλια ακριβώς γιατί φοβούνται αυτήν την κατάληξη. Φοβούνται να τους πάνε στα δικαστήρια. Και τι γίνεται με την προστασία των δικαιωμάτων. Πώς αυτά επηρεάζουν την διανομή μιας ταινία. Στη Γαλλία η περίοδος προστασίας ε, μιας ε, ταινία είναι πέντε χρόνια όταν έχει λάβει κρατική ε, χρηματοδότηση. Πέντε χρόνια από την ημερομηνία προβολή μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η ταινία αυτή διαθέσιμη σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά. Άλλη ερώτηση. η τσεχική βιομηχανία κινηματογράφου, η ιταλική, η γερμανική, το στούντιο Babelsberg, ε, αυτές οι μορφές καλύπτονται από κάποια πολιτική που θα έχει κάποια ωφέλη ή όχι στις ε, ίδιες τις παραγωγές. Έπειτα μας αναφέρεται αυτό το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται και οι φοροαπαλλαγές τις οποίες ε, απολαμβάνουν οι επενδυτές στις Ηνωμένε Πολιτείες. Διότι από όσο γνωρίζω, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιούν και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις και για το ότι μάλλον από ό,τι φαίνεται διαβάστερη μελέτη. Πρώτον, εμείς δεν κοιτάξαμε τι συμβαίνει με τις ε, παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις. Αυτό δεν ε, μας είχε ζητηθεί. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου απέναντί μου, οι οποίοι έχουν αναλύσει τα οικονομικά ζητήματα της ε, κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι φορά τη δεύτερη ερώτησή σας, εξετάσαμε τις ε, περίοδους προστασίας που αναφέρατε και εδώ πέρα αυτό έχει να κάνει και με την ευελιξία. Η περίοδος προστασίας είναι κάτι που αφαιρεί τη δυνατότητα ευελιξίας από τους παραγωγούς. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα να περάσουν σε ε, προσύμφωνα ε, ψηφιακή διανομή ε, όταν παρέλθε αυτή η περίοδος των πέντε ετών. Αυτό λοιπόν επιφέρει περιορισμούς στους παραγωγούς. Για παράδειγμα, όταν μια ταινία ε, έχει αυτούς τους περιορισμούς, ε, δεν μπορεί ούτε να πάει σε φεστιβάλ, ε, ούτε να προβληθεί αρκετά αν πρώτα δεν έχει ξεκινήσει η προβλήση Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελευταία ερώτησή σα, η απάντηση είναι όχι, μονολεκτικά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το 2014. Είναι η τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε στοιχεία σχετικά με τι άμεσε ενισχύσει. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για διάφορα έμεσα συστήματα, προγράμματα φοροαπαλλαγής ή ευνοϊκά δάνεια. Τα δάνεια βέβαια αυτά να σημειώσουμε ότι σπάνια αποπληρώνονται. Επομένως λοιπόν ε, δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα ε, πραγματικά ποσά. Δύο λοιπόν ε, από τις ερωτήσεις σας απαντήθηκαν. Δεν κατάλαβα όμως το τρίτο το ερώτημα και γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Αν δεν κάνω λάθος αφορά τη φορολογική πολιτική. Κι εγώ μόνο αυτό κατάλαβα από την ερώτηση. Μήπως θα μπορούσατε να την επαναδιατυπώσετε. Αυτό που εννοώ δηλαδή είναι η πολιτική στήριξη για ε, διάφορα στούντιο παραγωγής, όπως το Babelsberg. Υπάρχουν έξι κέντρα παραγωγής τέτοιου τύπου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εσείς ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή, την ε, στήριξη, τεχνική στήριξη και άλλη, ε, τι κάνετε. Το στούντιο Μπάμπελσπεργκ, από όσο γνωρίζω, είχε περάσει μία κρίση ε, στα κέντρα παραγωγής στην Ιταλία και την Τσεχία. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να απαντήσει. Τι γίνεται δηλαδή με τις κρατικές ενισχύσεις σε αυτά τα στούντιο παραγωγής, το, την Τσινετσιτά, το Μπάμπελσπεργκ ή στην ε, Τσεχία. Αν υπάρχουν δηλαδή κάποιες κρατικές ενισχύσεις ανεξάρτητα από επιμέρους ε, παραγωγές. Αν... Ναι, και ούτε αυτό είναι κομμάτι της μελέτης. Εμείς κοιτάξαμε γενικότερα τα φορολογικά κίνητρα για τη χρηματοδότηση ταινιών. Αυτή η ερώτηση λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν είμαι ειδικευμένος νομικός σε θέματα φορολογικού δικαίου και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να σας απαντήσω με σαφήνεια σε αυτό το ερώτημα. Αν όμως μας στείλετε γραπτά την ερώτησή σας, ίσως μπορέσουμε να την κοιτάξουμε να σας απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε με 4,20 ευρώ κατά κεφαλή είναι δύσκολο να ανοίξουν οι όταν ε, τόσες χιλιάδες αμερικανικά, αμερικανικές ταινίες ε, μπαίνουν στην χώρη αγορά. Αναφέρατε πάρα πολλούς λόγους, ε, παίρνουν χάρη ότι έχουμε υπερβολικές παραγωγές. Ε, ένα μέρος της, των γαλλόφωνων ταινιών ε, είναι 1% στο Βέλγιο και ε, η, ίδια, ο ίδιος ο οργανισμός ε, παραγωγής έκρινε καταθλιπτικές αυτές τις ταινίε. και δυστυχώς πολλές φορές μόνο στο φεστιβάλ των Κανών πηγαίνουν οι ταινίε αυτές. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή μια ταινία και έφευγαν οι θεατές από την αίθουσα είχα σμουριόνταν κατά τη διάρκεια της προβολής της είναι ένα μέρος του προβλήματος για τη Γερμανία. Υπογραμμίσατε ότι το νέο νομοθετικό ε, πλαίσιο ε, κυρίως ε, προωθεί την ποιότητα παρά την ποσότητα. Λιγότερε ταινίε, καλύτερης ποιότητα, Δηλαδή, το λαϊκό κινηματογράφο, τι θα το κάνουμε. Εμείς θέλουμε τελικά να εγκαταλείψουμε από ό,τι φαίνεται τις ποιοτικέ ταινίε και δυστυχώ να αντιγράψουμε τρίο στον Αμερικανικό κινηματογράφο. Πίτσε. Σας ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. I, didn't really detect the question. Ε, δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα σωστά το ερώτημα, αλλά ίσως ο συνάδελφος ο κ. Πόρτο θα μπορούσε να απαντήσει. Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως ε, ότι δεν ε, θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα πρέπει να είναι όπως οι αμερικανικές. Αυτό δεν είναι δική μα απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί. Απλώ λέμε πώς θα πρέπει να επανακαθορίσουμε την αγορά των ευρωπαϊκών ταινιών έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή γιατί ε, με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτό υπονομεύονται. Δεν λαμβάνουν δηλαδή ε, την προσοχή ε, που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε. Δεν λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν αμερικανικές. Απλώς τίθεται εδώ το ερώτημα του αν πώς προσεγγίζουμε την αγορά, αν την αντιμετωπίζουμε ως αγορά ή αν την αντιμετωπίζουμε ως τέχνη. Ε, πρόκειται δηλαδή εδώ για ε, με ασύμιξα αν θέλετε τμήματων κλάδων αγοράς και κλάδων τέχνης. Οπότε εδώ τίθεται το ερώτημα του τι ακριβώς εμείς επιθυμούμε ως κοινωνία, ως Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαντροβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και για την έρευνα. Υπάρχουν σαφή δεδομένα, αλλά κυρίως ποσοτικά. Ίσως αν υπήρχαν και ποιοτικά στοιχεία, τότε η παρουσία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σε σχέση με την ε, αρχή που αναφέρατε, την ε, γλωσσική αποκλειστικότητα. Είπατε ότι θα ήταν καλύτερη στη σύστασή σας. Θα ήθελα να αποσαφηνήσω. Πιστεύετε ότι η εδαφική αρχή αποτελεί την αιτία που θέτει εμπόδια και έχουμε λιγότερους θεατές, αν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά, η εδαφική αρχή αποτελεί την αιτία λιγότερων θεατών. Δεν είμαι σίγουρη αν η γλωσσική αποκλειστικότητα, αν εφαρμόσουμε τη δική σας σύσταση, θα μας οδηγούσε σε καλύτερα αποτελέσματα για να αυξήσουμε το κοινό και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των πολιτών στις ταινίε. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτή είναι η ερώτησή μου. Αυτή είναι η δική σας σύσταση, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά. Thank you very Σας δέχτε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα και για τα ευγενικά σας ε, σχόλια. Το ερώτημά σας ουσιαστικά είναι το εξής. Γιατί είμαστε υπέρ αυτού του μοντέλου της εκλογικής αποκλειστικότητας ε, και ποια προβλήματα θα επέλεγε. Η απάντηση είναι ότι δεν λέμε μέσα στην έκθεσή μας ότι αυτός ο χαρακτήρας της εδαφικής αποκλειστικότητας αποτελεί το βασικό πρόβλημα, την μητέρα αν θέλετε όλων των προβλημάτων για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι η εδαφική αποκλειστικότητα χρησιμοποιείται ως ε, σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση χρηματοδοτικού κεφαλαίου από την αγορά μέσω ακριβώς της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων προβολή στου παραγωγού που εργάζονται εντό τη επικράτεια ενό συγκεκριμένου κράτου μέλου. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ανέκαθεν η ευρωπαϊκή αγορά. Ε, και με τον οποίο, το οποίο μοντέλο εφήρμοζε πάντοτε ο κλάδο. Εμεί δεν ασκούμε κριτική σε αυτό το μοντέλο, απλώ αναφέρουμε ότι ενδεχομένω να μην είναι βιώσιμο το εν λόγω μοντέλο ε, ενώπιον ακριβώς ενός μέλλοντος όπου γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο ξεφεύγει από την αρχή αν θέλετε αυτής της ε, αυτό είναι το, το ζήτημα αν θέλετε η προβληματική που θίγει η έκθεσή μας. Και αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε εναλλακτικά μοντέλα τα οποία για παράδειγμα προτείνουν ακριβώς την, δημιουργία, την, την γλωσσικών ζωνών ή σημείων αποκλειστικότητας, αν θέλετε γλωσσικής αποκλειστικότητας, αντί για ε, εδαφική αποκλειστικότητα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού η εν λόγω αγορά ε, υποστηρίζει και μάλιστα εμφατικά τις πολιτισμικές ε, διαφορές. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι δοκιμάστε αυτό το εναλλακτικό μοντέλο. Είναι δηλαδή από οικονομική άποψη ένα βιώσιμο μοντέλο και ταυτόχρονα ε, έχει περισσότερο νόημα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα σε σύγκριση με το μοντέλο της διδαυτικής ε, αποκλειστικότητας. Εκτός βέβαια και αν αποφασίσουμε ότι θα επαναχωρήσουμε από το ευρωπαϊκό όρημα. τότε θα λύναμε το εν λόγω πρόβλημα, αλλά προφανώς δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, είμαι υπέρ της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση μου. Ευχαριστούμε. Ε, το λόγο έχει και πάλι η κυρία Τρούπελ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω λίγο σε ένα σε μία από τις βασικές της ε, θέσεις, ότι δηλαδή η νομοθεσία απομακρύνεται ένα και περισσότερο από την ε, εδαφικότητα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τα σχετικά μοντέλα αυτό το ζήτημα το συζητάμε εδώ και χρόνια ε, και το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα κάνουμε με την αγγλική γλώσσα. Εάν θεωρήσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κατανοήσουν την αγγλική γλώσσα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τις, γλώσσες, ε, για τις ταινίες σε αγγλική γλώσσα και τι σημαίνει για ταινίε, για παράδειγμα, στην πορτογαλική γλώσσα, γενικότερα για ταινίε σε ε, γλώσσες που μιλούνται από χαμηλό αριθμό άτομα. Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο λοιπόν για, την ευρωπαϊκή, για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Σε σύγκριση και σε σχέση πάντοτε με αυτή την απομάκρυνση που μας λέτε ότι λαμβάνει η χώρα από το μοντέλο της ε, ε, δαφικότητας. Ε, και να σας πω ότι στο πλαίσιο της ενισέας αγοράς παρόλα αυτά ο πολιτισμός είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ισχύουν και δεν θα πρέπει να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνε όπω αυτοί ισχύουν για παράδειγμα για τον κλάδο τη αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά τον τομέα του πολιτισμού. Και γνωρίζετε και έχει αναφερθεί αυτό και από τον σχετικό οργανισμό, τον Γαλλικό, ε, για τον πολιτισμό, ε, ότι έχει συγκεκριμένε ιδιαιτερότητε ο, ο ε, τομέα του πολιτισμού. Ειδικότερα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το geo-blocking είναι πολύ πιο προσεκτική και εκείνη σε σχέση πάντοτε με τον κινηματογράφο και ε, ο στόχος εδώ είναι να απαλλαγούμε από το geo και γενικότερα τα σύνορα. Αλλά Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, δηλαδή να καταργήσουμε το geo να κινηθούμε ε, προς αυτή την κατεύθυνση, μόνο εφόσον έχουμε δημιουργήσει εναλλακτικά και βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης. Και για να το επιτύχουμε αυτό, για να υπάρξουν τέτοιου είδου μοντέλα, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια θα πρέπει να επιληθεί και το ζήτημα του ποιο θα λαμβάνει αυτέ τι αποφάσει, δηλαδή τη παραγωγή λιγότερων ταινιών με υψηλότερο budget, με υψηλότερο προπολογισμό. Ε, ε, πράγμα βέβαια το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο όπω μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημά μου. Δηλαδή αυτή η γλωσσική αποκλειστικότητα που προτείνετε εσεί στην έκθεσή σας, τι ακριβώ θα σήμαινε αν εφαρμοζόταν στην πράξη. Λοιπόν, επειδή είναι συνδεδεμένα τα θέματα αυτά εγώ ήθελα να προσθέσω ότι εσείς δεν απαντήσατε στις αρχικές μου ερωτήσεις. Ε, ήταν ακριβώς αυτή η ερώτησή μου. Τι γίνεται με την γλωσσική αποκλειστικότητα όταν μιλάμε για μικρές χώρες. Δεν απαντήσατε και δεν απαντήσατε και στην ερώτηση το πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τις οποίες η συμβατική ελευθερία να είναι εντός ενός πλαισίου όπου δεν θα υπάρχουν ε, δυσανάλογα βάρη. Σκέφτομαι παραδείγματο χάρη τι μεγάλε πλατφόρμες ε, των γιγάντων του δικτύου και εκεί δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμβατική ελευθερία. Δηλαδή, εδώ ε, μιλάμε για τις επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα. Με συγχωρείτε που ξαναθέτω τις ερωτήσεις, αλλά δεν απαντήσατε. Καταρχήν να απαντήσω μία από τις ε, ερωτήσεις της κυρία Τρούπελ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και για την ε, πρόσθετη ερώτησή σας. Φυσικά, οι ταινίε μυθοπλασία ε, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο λέμε. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ καλή λόγη για ειδική μεταχείριση των ταινιών και φυσικά αυτό συμβαίνει σε αρκετού ε, τομεί που αναφέρατε ήδη. Αλλά επίσης ότι μάλλον θα είναι αγαθό να περιμένουμε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρη εδαφικότητα μακροπρόθεσμα και δεν το βλέπουμε αυτό με μια σειρά μέσων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε λύσεις που να καλύπτουν τις ειδικέ ανάγκες ε, αυτής ε, της ε, πολιτιστικής δημιουργίας, των ταινιών δηλαδή, χωρίς να αγνοούμε τις, ε, τα μεγαλύτερα αιτήματα της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή ισχύει. ισχύουν οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς ακόμη και για τις ταινίε. Έτσι λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει δύο λύσεις. Δηλαδή, όχι απλώς να εγκαταλείψουμε την εδαφικότητα και να έχουμε γλωσσική αποκλειστικότητα που δεν είναι καθόλου επαναστατική. Ήδη συμβαίνει στην πραγματικότητα σε πολλές αγορές γιατί έχουμε επικάλυψη πολλών εδαφικών επικρατιών ως προς τη γλώσσα. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Σε κάποιες περιοχές δεν είναι επαναστατικό λοιπόν και επίσης αυτό ανασωποιεί την, τον κλάδο του κινηματογράφου από τον ε, από το δίκαιο του ανταγωνισμού, δηλαδή να έχουμε ε, ουσιαστικά ε, προστασία του κινηματογράφου από το δίκαιο ανταγωνισμού. Και εσείς και η κυρία Κώστα θέσατε μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το τι σημαίνει μία μετακίνηση προς τη γλωσσική αποκλειστικότητα για τις μικρές γλώσσες στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο Γιος Σπορτ μπορεί να απαντήσει καλύτερα στην ερώτηση αυτή από μένα και του δίνω το λόγο. Πιστεύουμε ότι δεν θα άλλαζαν πολλά στην πραγματικότητα, γιατί σήμερα παράγονται ε, ταινίε από μικρότερε χώρε και βλέπουμε ότι οι μικρότερε χώρε παράγουν περισσότερε ταινίε τα κεφαλή από τι μεγαλύτερε χώρε και δεν υπάρχει κανένα λόγο να άλλαζε αυτό αν αλλάζατε το μοντέλο χρηματοδότηση ε, προ ένα μοντέλο που θα βασιζόταν στην γλωσσική αποκλειστικότητα. Το πιο βιαστικό ερώτημα είναι τι θα γινόταν στι αγγλόφωνε ταινίε και το αναφέρατε αυτό. Αν προσπαθείτε να δείτε το μέλλον, μπορεί να περιμένετε ότι η άδεια της αγγλικής εδοχής σε ένα τέτοιο ε, μοντέλο άδεια θα αξίζει περισσότερο και θα γινόταν ε, κάτι πιο πολύτιμο ακόμη, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα σε κάθε χώρα που ε, ουσιαστικά είναι ικανοποιημένη μόνο αν έχει πρόσβαση στην αγγλική εκδοχή, δεν χρειάζεται υπότιτλους, ε, ούτε μεταγλώτηση. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι μικρή αυτή η ομάδα και αν δείτε τους οικονομικούς μηχανισμούς από πίσω δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο λόγω του Brexit, <clears throat> αλλά επειδή Σήμερα το εισόδημα κατά κεφαλή στις χώρες όπου μητρική είναι τα αγγλικά είναι αρκετά υψηλό στο ευρωπαϊκό τοπίο. Ήδη λοιπόν έχουμε μία άδεια που κοστίζει περισσότερο. Είναι πιο πολύτιμη από τη άδεια στην Πορτογαλία ή στη Λετωνία. Αν το δείτε από τη σκοπιά της αγοράς, το γεγονός ότι θα υπάρχει κάποια διαρροή για να το πούμε έτσι, τη αγγλική εκδοχή ταινία προς ε, αγγλόφωνους πληθυσμούς αλλά μέλη δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα για τη χρηματοδότηση των ταινιών. Έτσι αναλύουμε το θέμα αυτό και όπως σας είπα για τις μικρότερες ε, χώρες και τις μικρότερες γλώσσες δεν θα άλλαζαν και πολλά στο μοντέλο αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. και του προσκεκλημένου και τους ε, συναδέλφου για αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πολύ για τη συζήτηση και στο σημείο αυτό μπορούμε να κλείσουμε το σημείο 8, 7 της ημερήσιας διάταξης. Térjünk rá a következő pontunkra. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της σας διάταξης. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης που αφορά την πρόταση αποφάσης του Συμβουλίου με την οποία εξοδοτούνται τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, προστασία και παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Η συγγήτρια είναι η Έμα Μακλάρκιν. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 24 Μαρτίου 12 ώρα το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στη συνέχεια και η γνωμοδότηση αυτή είναι πάνω στην έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία θα ψηφίσει στις 18 Φεβρουαρίου. Η συγγήτρια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι η Σίλβια Κάουφμαν και αποφασίσαμε λοιπόν να εργαστούμε γρήγορα έτσι ώστε μέχρι να ψηφίσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εμείς να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να εργαστούμε στην αγγλική γλώσσα. Η γνωμοδότηση αυτή βρίσκεται στο στάδιο της ε, έγκρισης, της ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε με ναι ή όχι. Η Τροπολογίες λοιπόν μπορούν να κατατεθούν μόνο γραπτός και θα γίνουν παραδεκτές μόνο εάν γίνουν δεκτές και από την εισηγήτρια. Η γραμματεία λοιπόν θα σας στείλει σχετική ενημέρωση που θα εξηγεί πώς ακριβώς ε, θα ε, γίνει αυτή η διαδικασία των συστάσεων. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στους ε, συναδέλφους. Έχετε το λόγο κύριε Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ασφάλεια στους αθλητικούς αγώνες είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για το προσωπικό που εργάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να μην φοβούνται βίες εκρήξεις και περιστατικά μέσα ε, σε ένα αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιωθεί η ασφάλεια και μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί και η γενικότερη ατμόσφαιρα σε έναν ε, χώρο, σε ένα στάδιο. Αυτό θα ωφελήσει και τη διεξαγωγή των αγώνων. Για παράδειγμα, η Premier League της Αγγλίας κατάφερε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του χουλικανισμού ε, μόλις πρόσφατα, το οποίο ήταν πραγματική αρρώστια ε, την δεκαετία του 80 με αποκορύφωμα τα επεισόδια του 1985 στον αγώνα liverpool liverpool-juventus εδώ στις Βρυξέλλες. Η το αποτέλεσμα αυτών των ε, γεγονότων μετά τον ε, διαχωρισμό ε, των φιλάθλων σε δύο ομάδες ήταν να στριμωχτούν σε έναν τοίχο ο οποίος στη συνέχεια κατέρευσε με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Ως αποτέλεσμα αυτών των επεισοδίων, το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1985 δημοσίευσε ένα, μια συμφωνία η οποία τέθησε ισχύ έξι μήνες αργότερα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς στους ποδοσφαιρικούς και άλλους αθλητικούς αγώνες για την ε, πρόληψη βίας. Ο κανονισμός αυτός απέτησε διεθνή συνεργασία και δημιουργήθηκε μία μόνιμη επιτροπή η οποία παρακολουθούσε την εφαρμογή της ε, συμφωνία αυτή, Αποτελούταν από εμπειρογνώμονε του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλους εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη, αρμόδιες αρχές και της, ε, την Ίντερπολ και τις ε, αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Όμως ο κανονισμός αυτός είναι πλέον παροχημένος, χρειάζεται αναθεώρηση της συμφωνίας, γι' αυτό και συζητούμε σήμερα το θέμα αυτό εδώ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του έτσι ώστε το Συμβούλιο να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη προσέγγιση στους ε, αθλητικούς αγώνες. Χρειάζεται μια πολυτομεακή προσέγγιση, άριστη συνεργασία έτσι ώστε το ποδόσφαιρο και άλλοι, άλλες μορφές αθλητισμού να ξαναγίνουν ασφαλείς για όλους. Αυτό προϋποθέτει ασφάλεια των ε, υπηρεσιών και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν επικαλύψεις. Γι' αυτό χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και όχι μόνο από έναν ε, οργανισμό, διοργανική συνεργασία. Το Συμβούλιο της Ευρώπη λοιπόν και τα κράτη-μέλη είναι τα αρμόδια που θα αποφασίσουν. Η μόνη προπόθεση για τα κράτη-μέλη είναι η δημιουργία ενός ε, σημείου, ενιαίου σημείου επαφής ε, και ανταλλαγή πληροφοριών ε, ανάμεσα στι αρχές και στα κράτη-μέλη για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην έκθεσή μου, στη γνωμοδότησή μου μάλλον για την έκθεση της Επιτροπής Ελίμπε, συστήνω να δώσω το Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του. Είναι προ όφελο της ασφάλειας να διευρυνθούν οι ε, κανόνες και να επικαιροποιηθούν να επικαιροποιηθεί μάλλον η συμφωνία η οποία θα πρέπει να προποθέτει σύγχρονες ε, υποδομές. Υπάρχει, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, κάποιες βέλτιστες πρακτικές από τα κράτη-μέλη που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Για παράδειγμα, ε, η περίπτωση της Γερμανίας με την ασφάλεια στις ε, θέσεις όρθιων. Ζητώ λοιπόν στη γνωμοδότηση την συμφωνία των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να συνεχίσει να αποτελεί η ασφάλεια στους αθλητικούς αγώνες ε, ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο κύριος Ζαγοράκης, ο οποίος απουσιάζει, δεν θα τον αντικαταστήσει κάποιος. Πολύ ωραία, μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες δεν είναι εδώ επίσης. Αποουσιάζει ο σκιώδης εισηγητής. Δεν βλέπω κανέναν σκιώδη εισηγητή. Άρα λοιπόν όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει το λόγο από τους υπόλοιπους. Παρακαλώ εσείς. Κυρία Μπίλντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ήδη η σύμβαση έχει κυρωθεί επί της ουσίας από την Γαλλία, όμως τίνει να προσεγγίσει το θέμα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των αγώνων μαζί με τους συνδέσμους ε, στη Γαλλία ε, από το 2011 και βάσει της νομοθεσία του 2016 ελέγχονται οι σύνδεσμοι. Το βλέπουμε ε, στη Γαλλία και στο Ερμένο Βασίλειο ότι υπάρχουν τεράστιες διοικητικές απαγορεύσεις. Όμως ποια είναι αυτή που βιοπραγούν όταν ε, υπάρχει βία. Συχνά έχουμε μία μικρή μειοψηφία που δεν ανήκουν ε, στον κόσμο ε, του ποδεσφαίρου και υπάρχει και η απειλή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ε, το να στιγματίζουμε τους οπαδούς ε, ως ε, πιθανούς χούλιγκαν ενώ είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου μου φαίνεται άδικο και αντιπαραγωγικό. Γι' αυτό εγώ ε, συμφωνώ με κάθε πρόταση που θέλει να αποδώσει τον συντροφικό χαρακτήρα σε αυτό το σπορ. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νέκοβ είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Καλημέρα συνάδελφοι. Ζήτω συγγνώμη για την αργοπορία. Θα ήθελα λοιπόν να πω πως η συμφωνία αυτή είναι μια νομικά δεσμευτική πράξη η οποία καθιστά υποχρεωτική τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλόμενα μέρη. Η συμφωνία λοιπόν αυτή 120.985 υποτέθησε ισχύ μετά την τραγωδία του Χέισελ όπου 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους χρειάζεται επικαιροποίηση έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, σύγχρονες προκλήσεις. Τρεις είναι αυτές. Ασφάλεια, ασφάλεια στους ε, χώρους αγώνων, έτσι ώστε οι αγώνες να διεξάγονται με επιτυχία χωρίς προβλήματα. Τα κράτη-μέλη δεν είναι τα μόνα υπεύθυνα γι' αυτό. Όλοι οι οργανισμοί, οι φορείς ε, των αγώνων και φυσικά το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αρμόδιο για την ε, εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Το Erasmus Plus επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία τέτοια προσέγγιση έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η βία. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόκληση και όχι τόσο στο μετά αφού έχουν σημειωθεί βία επεισόδια. Θεωρώ επίσης πως θα πρέπει να στηρίξουμε ως Κοινοβούλιο τη συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διακόνου έχει το λόγο. Και κύριε κυρία Κώστα. Εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές για αυτή τη σημαντική αναθεώρηση της ε, σύμβασης. Ε, πρέπει να πω ότι είναι λυπηρό να μιλάμε για τον αθλητισμό και να το συνδέουμε πάντα με τη βία, για κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και τη ζωή των ε, ατόμων. Και αυτό δυστυχώς προδίδει την αξία του αθλητισμού και συνδέεται το ποδόσφαιρο με τέτοιες αξιολογήσεις και θα πρέπει να μας οδηγήσει αυτό στο να σκεφτούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εμπορική και η κανονική διάσταση του ποδοσφαίρου και δυστυχώς ε, ε, ουσιαστικά αποδυναμώνεται το ίδιο το ποδόσφαιρο και ε, βλέπουμε τι γίνεται και με τους χούλιγκαν και στην Ιταλία έχουμε πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια και δυστυχώς ε, έχουμε πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις άλλες φύσεις που βρίσκουν την ευκαιρία να μπορέσουν ε, να εκφράσουν με βίαιο τρόπο τη στάση τους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Εδώ προσπαθούμε να αναφερθούμε σε κάτι που θεωρείται παράδεκτο στη ρίζα του. Τώρα, εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα στην ε, αναθεώρηση, ότι πάμε πέρα από το θέμα της ε, συνεργασίας ε, Εδώ βασιζόμαστε ε, στο άρθρο 185 της συνθήκης και είναι σημαντικό να το μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να δούμε και πώς γίνεται ο σχεδιασμός και η διαχείριση και η συμμόρφωση με τους ε, κανόνες ε, σε ό,τι αφορά και την οργάνωση εντών των σταδίων αλλά και σε ό,τι αφορά την παρέμβαση, τη μεθοδολογία επέμβασης αλλά και πρόληψη. Σκέφτομαι, παραδείγματο χάρη, ότι παντού θα πρέπει να υπάρχουν κάμερε για να μπορούμε να ελέγχουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστε που προβαίνουν σε βιοπραγίε. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι να προβλέψουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορα στάδια. Δηλαδή έχουμε ε, το θέμα της διαχείρισης, το θέμα της ασφάλειας ε, και το θέμα της ευθύνης των αθλητικών ε, ενώσεων. Δεν αναφερόμαστε πολύ σε αυτό, όμως είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε στο νου μας και για το μέλλον. Και ευχαριστώ και πάλι την συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διακόνου τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα μεγάλος ε, οπαδός του ποδοσφαίρου, ούτε ιδιαίτερα αθλητικός τύπος, ε, όμως παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή τι συμβαίνει και βρισκόμαστε ενώπιον ενός φαινομένου που ξεκίνησε καταρχήν ε, μεμονωμένα, βλέπαμε τους χούλιγκαν στην Αγγλία και όλο αυτό το βλέπαμε εξ αλλά σιγά σιγά διαδόθηκε το φαινόμενο αυτό και άρχισε να εμφανίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν ε, αρκεί να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο μόνο σε σχέση με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γιατί κάποια στιγμή και το είδαμε αυτό όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά και στη χώρα μου, όταν κάποιοι άνθρωποι σε δημόσιο χώρο ε, ζητούν ε, ε, την άδεια να κάνουν μια διαδήλωση, να εκφράσουν την άποψή τους. Πολύ ωραία τη μια μέρα, τη δεύτερη μέρα, όμως κάποια στιγμή εμφανίζεται μια μάζα βίαιων ανθρώπων που αλλάζουν την όλη κατάσταση και βλέπουμε να γίνεται ξαφνικά της τρελής. Και οι άνθρωποι αυτοί αγνοούν, παίρνουν το σχάρι, ε, την αιτία της διαδήλωσης, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έρθουν σε συγκρούσεις με τους αστυνομικούς. Δηλαδή τους ενδιαφέρει η βία για τη βία, τέχνη για την τέχνη όπως λέμε. Και είναι αλήθεια ότι σε κάθε συλλογικότητα υπάρχει ε, ένας πυρήνας τέτοιων ομάδων που ε, μπορεί το χάρη να είναι και βίοι στην ίδια την οικογένειά τους ή στο δρόμο. Ε, τέλος πάντων, με την ευκαιρία αυτή αρχίζουν να συγκεντρώνονται, να μαζεύονται και να γίνονται βίαιοι σε ομάδα, στην ομάδα. Δηλαδή το θέμα είναι ε, ότι έχουμε εδώ συλλογική ευθύνη και όχι μεμονωμένη. Γιατί, παραδείγματο χάρη, μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιε κάμερε και να εντοπίζονται κάποιοι πιθανώ ε, βίαιοι άνθρωποι. Αυτό δεν αρκεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά δρούν ε, κάπως υπερβάλλω, αλλά σαν να είναι παραστρατιωτικές ομάδες. Και ουσιαστικά προετοιμάζονται και με την ευκαιρία αυτή ε, ουσιαστικά το εξασκούν. Μόνο και μόνο για να έρθουν σε συγκρούσεις. Είναι δηλαδή πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, κατά την άποψή μου, αναπτύσσεται και εμφανίζεται και σε περιοχές όπου δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται, όχι μόνο, παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο, Μπορούμε να το δούμε, παραδείγματο χάρη, σε κάποιε ε, συλλογικέ διαμαρτυρίε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει το φαινόμενο αυτό να το δούμε μέσω των υφιστάμενων ενώσεων. Θα πρέπει την ευθύνη να την αναλάβουν οι σύνδεσμοι ενώσεις καταρχήν και στη συνέχεια τα άτομα. Μπορεί να εργαστεί κάποιο με τι ενώσει, ε, μπορεί να τιμωρηθούν οι ενώσει, οι σύνδεσμοι, να του επιβληθούν κυρώσει, ε, να τύχουν απαγόρευση κτλ. Επομένω, είναι πολύ επικίνδυνο το φαινόμενο και θα ήθελα να του προσδώσουμε και την απαραίτητη προσοχή γιατί γίνεται όλο ένα και πιο σοβαρό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Φέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εξαιρετική κυρία Πρόεδρε, να πω ότι υποστηρίζω και εγώ την αλλαγή της ενόγου συμφωνίας και υπόσχομαι στην εισηγήτρια ότι θα έχει τη δική μου υποστήριξη και θα συνεργαστώ και με τους υπολείπους ε, σκιώτησε εγώ θυμάμαι τα όσα συνέβησαν τότε στο Βέλγιο πριν από 3,5 δεκαετίες και το πόσα πολλά ε, θύματα ε, είχαμε ε, μετά από αυτήν την σύγκρουση μεταξύ των δύο διαφορετικών ομάδων φιλάθλων. Αλλά βέβαια εκείνο το γεγονό αποτελέσε και ένα σημείο καμπή. Γιατί έκτοτε και η δική μου χώρα και μια σειρά από περαιτέρω χώρε άρχισαν να ασχολούνται πλέον εντατικότερα με αυτό το φαινόμενο. Ε, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο ε, κατάφερε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα με αποτέλεσμα να μην είναι ε, πλέον απαραίτητο το να υπάρχουν κάγκελα στα διαφορετικά γήπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που αποτελούσε ένα κανονικό, αν θέλετε, εξοπλισμό για τέτοιους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και το υπόδειγμα που έδωσε λοιπόν, που δημιούργησε αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα παράδειγμα που ακολούθησαν και μια σειρά από άλλες χώρες και διαπιστώνουμε ότι μία σειρά από χώρε οι οποίε αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα βία σε ό,τι αφορά την διοργάνωση αθλητικών ε, αγώνων, δεν τα αντιμετωπίζουν πλέον στον ίδιο βαθμό. Τόσο εντό τη Ευρώπη όσο και εκτό. Ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον μπορεί να αυλυνθεί λίγο το εν λόγω πρόβλημα γιατί βέβαια συχνά συνοδεύεται η αύξηση της βίας σε τέτοιου είδους αγώνες από ε, αντίστοιχες ε, κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις. Εφόσον όμως λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ναι, είναι δυνατόν να μειωθεί, να μετριαστεί η βία. η ιστορία των διαφόρων ε, φιλάθλων αν θέλετε, ε, του ποδοσφαίρου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ε, αυτό αφορά και την πρώην Ιουκοσλαβία. Δηλαδή κάθε φορά όπου είχαμε δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες είχαν μια αναμέτρηση μεταξύ τους δημιουργούνταν αυτομάτως τέτοιου είδους ε, ομάδες φιλάθλων, ουσιαστικά χούλιγκαν, δηλαδή που είχαν τάσεις βίας. Ε, και αυτό που συνέβαινε στην ε, πρώην Ιουκοσλαβία είναι η ε, μία ομάδα φιλάθλων, από τη μία δηλαδή ομάδα να παρακολουθείται από την πολιτική μυστική αστυνομία, ενώ η άλλη ομάδα να παρακολουθείται από την στρατιωτική στην αστυνομία. Ε, βέβαια αυτό το μοντέλο στη συνέχεια μετεβλήθη, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό να πούμε εδώ είναι ότι η η ηγεσία των ελόγων ε, συνδέσμων ε, φιλάθλων ε, συμμετέχει σε όλες τις δράσεις από την πλευρά αυτών των φιλάθλων και εγώ έχω ασχοληθεί με την ιστορία των χούλιγκαν και πραγματικά θα πρέπει να πω ότι οι ηγέτες των εν λόγω ομάδων φιλάθλων ενσωματώθηκαν αν θέλετε μέσα στους ε, στις, ε, ε, στους συνδέσμους της ίδιας της ομάδας των φιλάθλων και άρχισαν να εδραιώνονται, να θεσμοθετούνται κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ομάδες των φιλάθλων απλώς και μόνο σε περιφερειακό φαινόμενο. Μπορούν να αποτελέσουν τμήμα της κανονικής ζωής, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή να αποτελούν τμήμα των ίδιων των αθλητικών οργανώσεων οι συνδέσμοι φιλάθλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι τώρα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εκπροσωπός της, θα ήθελα να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι από την Γενική Διεθνή Home ε, και εκπροσωπώ. Ε, ε λέγομαι Δημήτρη Αγιοτάκο. και να πω ότι από την πλευρά της Επιτροπής ε, εκτιμούμε πραγματικά την θετική στάση που έχει εδώ η συγκήτρια, κυρία Μακλάρκιν, και εκτιμούμε και τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν από την πλευρά των ε, στιωτών εισηγητών και των υπολείπων ε, ομιλητών σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Και ελπίζουμε πως και αντίστοιχη στάση θα τηρήσει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, στη ε, συνεδρίασή της 29 Ιανουαρίου και στις 18 Φεβρουαρίου στη συνέχεια, έτσι ώστε τελικά να λάβουμε την οριστική συνένεση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου από την πλευρά του Συμβουλίου να γίνει η υιοθέτηση και να επιταχυνθεί η διαδικασία της ε, κύρωσης εν λόγω σύμβασης από τα κράτη-μέλη, γιατί είναι που θα πρέπει να το κάνουν ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Η συγκήτρια έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για το ενδιαφέρον που δείχνετε ε, για αυτό το ζήτημα. Πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ε, ότι η φίλαθλοί μας ε, πραγματικά είναι ασφαλείς στα γήπεδά μας και πραγματικά σέβονται τους κανόνες που ισχύουν ε, εκεί. Δηλαδή, ας ε, κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν απάθος ε, για τον αθλητισμό να συνεχίσουν να το χαιρετούν. Ε, καθώς ε, αναλαμβάνω για τελευταία φορά ω εισηγήτρια εδώ στο Ευρωπαϊκό μα ε, Κοινοβούλιο, ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλους ε, για την ε, υποστήριξη και πραγματικά χαίρομαι που η τελευταία μου ε, νομοδότηση για την οποία είμαι αρμόδια αφορά αυτό το ζήτημα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου γιατί με ενδιαφέρει πολύ και πραγματικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σεβαστούμε και να τηρήσουμε τις σχετικές αξίες και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πραγματικά όλου για την υποστήριξή Σα Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω λοιπόν προς ενημερωσή σας ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 24 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών και στις 11 ακριβώς θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με την ε, συνεδρίασή μας ε, και με ιδιαίτερη μου χαρά θα ήθελα να παρουσιάσω τους εκπροσώπους της Ρουμανικής Προεδρία ε, σήμερα εδώ και συγκεκριμένα έχουμε την Υπουργό Εθνικής Επαιδείας κυρία Κατερίνα Ανδρονέσκου τον Υπουργό πολιτισμού και εθνικής ταυτότητας ε, τον κύριο Βαλέρ Ντάνιελ Μπράς και τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού τον κύριο Κωνσταντίν Μπογκδάν Ματέι. Σας ε, καλωσορίζω λοιπόν και τους τρεις υπουργούς ε, θερμά εδώ στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε το Brexit δημιουργεί μια σειρά από νέε προκλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια η δική σα Προεδρία είναι η οποία θα χρειαστεί να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, πράγμα το οποίο βέβαια δυσκολεύει το έργο σα. Επιπροσθέτω, έχετε και τι επόμενε εκλογέ του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου κατά την Προεδρία σα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσετε να ολοκληρώσετε όσο το, περισσότερο, ε, όσο το δυνατόν ε, περισσότερα νομοθετικά ζητήματα και να καταλήξετε σε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, σε αυτή την περίοδο. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά ε, το Εράσμους, ε, το Σώμα Αλληλεγγύης και ένα ακόμα ζήτημα η Επιτροπή υπέβαλε πολύ καθυστερημένα τις δικές της προτάσεις με αποτέλεσμα βέβαια να είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων μετά από την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ε, θεωρούμε πως θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στους δικούς μας τομείς, δηλαδή του πολιτισμού, του αθλητισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Οπότε θα ήθελα να δώσω σε εσά, στου τρει υπουργού, στον καθένα τον λόγο για 10 λεπτά, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνει και ένα γύρω συζήτηση με τα μέλη τη Επιτροπή μα. Ε, νομίζω πω η κυρία Αντρονέσκου θα είναι η πρώτη υπουργό που θα πάρει το λόγο. Έχετε λοιπόν τον λόγο, κυρία Αντρονέσκου, σα καλωσορίζω θερμά για 10 λεπτά. Σα ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι συμμετέχοντες, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας και να σας μιλήσω για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Ως καθηγήτρια καταρχήν θεωρώ ότι η παιδεία είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους και σίγουρα η παιδεία είναι ο τομέας που ενδυναμώνει τις ευρωπαϊκές αξίες και τη διαβίβαση των ευρωπαϊκών αξιών σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βεβαιότητα ότι μέσω της παιδείας μπορούμε να πετύχουμε τη συνοχή ως κοινή ευρωπαϊκή αξία. Σας μιλώ και ως Υπουργός Παιδείας αλλά και ως ε, ε, πρώην δικαιούχος των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων και από τη θέση αυτή χαίρομαι που μπορώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα σχέδια και τα προγράμματα που έχει εγκρίνει για τα, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι για τη Ρουμανία, αλλά και όχι μόνο, τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ήταν μια ανοιχτή οδός για την επικοινωνία και για τη συνεργασία. Μέσω αυτών των προγραμμάτων σας διαβεβαιώ από τη θεσμική μου θέση ως Πρίτανη, ως κοσμήτορας μπόρεσαν να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας. Αναπτύξαμε προγράμματα έρευνας με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προγράμματα μετευχιακών, είχαμε ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά για μας και επίσης κάτι πολύ σημαντικό ήταν και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων μέσω της οργάνωσης διδακτορικών θέσεων. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω ότι τα προγράμματα που θέτει στην Ρουμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου της παιδείας. Σίγουρα θα πρέπει να διαχειριστούμε φακέλους με πολύ μεγάλη ευθύνη και ανοιχτό πνεύμα. Ζητάμε τη δική σας υποστήριξη γιατί δεν πιστεύουμε ότι μόνο η Ρουμανία μπορεί να επιλύσει τα θέματα όλα αυτά, αλλά μόνο μέσω της συζήτησης μαζί σας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να καταλήξουμε στις κατάλληλες λύσεις και να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές ιδέες και αξίες τα συστήματα υψηλή ποιότητα ε, για την εκπαίδευση και ε, τη μέρημνα των παιδιών. Ανοίγουν ε, νέε οδού. Σήμερα οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση μιλούν για τη σημασία των γνωστικών δεξιοτήτων, απόκτησης γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τα προγράμματα αυτά αναπτύσσεται η δυνατότητα να ενταχθούν όλα τα παιδιά σε προγράμματα εκμάθησης και σε προγράμματα μέριμνας από τις πολύ μικρές ηλικίες. Στην Επιτροπή Παιδείας συζητείτε αυτό το πρόγραμμα. Ήδη υπήρξαν σχετικές συναντήσεις και ελπίζω ότι με τη δική σας βοήθεια των θεσμικών οργάνων θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο και να το ολοκληρώσουμε. Εμείς αυτό επιθυμούμε και βασιζόμαστε στη δική σας υποστήριξη. Ταυτόχρονα η πλήρης ε, προσέγγιση της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών αποτελεί μια οδό επικοινωνίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια οδό μέσω της οποίας οι νέες γενιές μπορούν ε, να συνονοηθούν και να συνεργαστούν πιο εύκολα και έτσι διασφαλίζεται και η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών καθώς ε, θα υπάρχουν πιο εύκολες και άμεσες συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς ε, είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα και επίσης ε, ελπίζουμε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτός, να υπάρχει αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος της δικής μας Προεδρίας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα αλλά και ιδιαίτερα πολύπλοκα ταυτόχρονα που αναμένουν με υπομονησία οι Ευρωπαίοι πολίτες και τουλάχιστον οι νέοι είναι σίγουρα το Erasmus Plus. Το πρόγραμμα Erasmus ήδη έχει επιφέρει θετικές ε, συνέπειες σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το μελλοντικό σχέδιο μέσω διάφορων προσθήκων που έχετε προτείνει εσείς ε, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και θα φέρει περισσότερα ωφέλη στους συμμετέχοντες. Αναφέρομαι εδώ φυσικά στην τυπική ή άτυπη μάθηση, αναφέρομαι στην κινητικότητα που οι νεότερες ή όχι τόσο νέες γενιές ε, θα ε, μπορούν να ελοποιήσουν μέσω αυτού του προγράμματος και στην αφομοίωση του πολιτισμού των ε, ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, αναφέρομαι στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα δίκτυα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Πιστεύω ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων το πρόγραμμα Εράσμους θα διευρύνει τον ευρωπαϊκό χώρο παιδείας. Να ήθελα να προσθέσω και ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Παιδείας αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη να προωθήσει τις αξίες της, μια ευκαιρία για μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη, για μια Ευρώπη όπου οι πολίτες θα έχουν ε, ίσα δικαιώματα και θα μπορούν να προωθήσουν ε, τις βασικές ε, δεξιότητές τους που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες ε, κατά την αναζήτηση επαγγελματικής διαδρομίας. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι εκπονήσατε τον κανονισμό του προγράμματος Εράσμους. Το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί ήδη σε πολλά εθνικά κοινοβούλια το Συμβούλιο δέχτηκε εν μέρη τη Γενική Συμφωνία για τον κανονισμό αυτό και αν κατορθώσουμε να έχουμε ένα ξεκάθαρο προπολογισμό για το πρόγραμμα Εράσμους, μπορεί να αυξηθεί και η πιθανότητα να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι και ίσως να υπάρχει και δυνατότητα ολοκλήρωσης αυτού του προγράμματος. Τώρα, η κινητοποίηση στην ε, κινητικό, της κινητικότητας των πανεπιστημίων στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι σημαντικό που προκύπτει και από την αυξημένη αποτελεσματικότητα του Εράσμους. Έχω την πεποίθηση ότι στις ε, συνεδριάσεις ε, του Βουκουρέστη, όπου σας ε, καλώ να παρευρεθείτε, και να γνωρίσετε τα προβλήματα που συζητάμε εμείς σε αυτές τις συνεδριάσεις, αλλά φυσικά σας καλούμε να γνωρίσετε και τη χώρα και τη Ρουμανία Αυτές οι συνεδριάσεις λοιπόν θα αποτελέσουν προσθεμένη αξία των προσπαθειών μας σε αυτό το σημαντικό τομέα συνεργασίας. Πριν να κλείσω θέλω να σας διαβεβαιώσω για μια φορά ακόμα για τη διαθεσιμότητα της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα πολύ σημαντικά θέματα της παιδείας. Ένας από τους μεγάλους ιστορικούς π.χ. η Ρουμανία και θα παρέθετα τον Νικολά Γιώργα, έλεγε «Η παιδεία είναι όλα όσα βλέπεις και όσα ακούς». Επομένως, είναι δικό μας καθήκον να στραφούμε στους νέους, προκειμένου να εκπαιδευτούν και να αφομοιώσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου επιτρέψατε να πω δύο λόγια από το βήμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τους συντονιστές, τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Για δύο λεπτά. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής. Κάπως έτσι θα γίνει, ερωτήσεις, απαντήσεις, έτσι να είναι πιο ζωντανά τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Σόιντροβα. Ποιο από εσά ε, θέλει το λόγο σήμερα, δεν ξέρω. Κυρία Σόντρεβα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, κυρία Υπουργέ. Για αυτό το εξάμεινο βλέπω ότι η προτεραιότητα είναι ο προπολογισμό για το πρόγραμμα Erasmus Plus. Για την χρονική περίοδο 2021-2027. Πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει προτείνει ένα καλό προϋπολογισμό, αλλά η δική μας Επιτροπή θα ήθελε ακόμη περισσότερα κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να διευρύνουμε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί το πρόγραμμα αυτό θα θέλαμε να μπορεί να περικλεί περισσότερους ανθρώπους να μπορούν να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι νέοι στο πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά αφορά κυρίως τον συνάδελφό σας που είναι αρμόδιος υπουργό για την νεολαία. Το, πρόγραμμα, το κοινό πρόγραμμα για την παιδεία, τον πολιτισμό και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα στην Επιτροπή μας, στην Ολομέλεια και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να υποστηρίξετε αυτό το πρόγραμμα στις ε, διαπραγματεύσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τους ε, νέους ηλικιακής ομάδας 18-30. Ε, και ελπίζουμε έτσι να προωθηθεί η ελληνική και ο θελαντισμός. Ελπίζω να σημειώσετε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κυρία Σόρτρεβα. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν ως ε, καθηγήτρια ε, Βεβαίω και θα υποστηρίζα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, έχουμε και τις εκλογέ και θα πρέπει να συζητήσουμε και το Brexit, αλλά εγώ φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σας και θα προσπαθήσω να υποστηρίξω την αύξηση του προπολογισμού για το Εράσμος. Αν το πετύχουμε αυτό, νομίζω ότι καταρχήν θα είναι δική σας επιτυχία και εγώ θα είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Αυτό θα το πετύχετε με τη δική σας ψήφο και βεβαίως εγώ θα σας υποστηρίξω στο πρόγραμμα αυτό γιατί συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι για τη νέα γενιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Σίλβια Κώστα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Εκτίμησα τα όσα είπατε για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ρουμανική Προεδρία. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Γιατί ουσιαστικά είναι και στην περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών. Και Ουσιαστικά θα πρέπει να βοηθήσετε και το Κοινοβούλιο να υιοθετηθούν ή να ολοκληρωθούν τουλάχιστον σημαντικές διαπραγματεύσεις. Είδα ότι μεταξύ των προτάσεων που υποβάλλετε θέλετε μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στο να υπάρχει ποιοτική εκπαίδευση και παιδεία για όλους τους νέους, κυρίως ε, Στου νέου με μικρότερε ευκαιρίε. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μα. Επίση, ζητήσατε ενίσχυση του προπολογισμού για το Εράσμους και να υπάρχει και νέα προσέγγιση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα αφορά τα δύο ψηφίσματα συστάσεις που εσείς θέλετε να υλοποιήσετε. Πιστεύω ότι το γλωσσικό θέμα αποτελεί ένα ιστορικό πρόγραμμα, πρόβλημα που ίσως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί καλύτερα, να έχουμε καλύτερε. Ε, πρακτικέ σε ό,τι αφορά τι ε, εθνοτικές μειονότητε, είναι ένα εκρηκτικό ζήτημα και το άλλο ζήτημα αφορά την ε, μεγαλύτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στην υπιακή ηλικία νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες ε, έρευνες ε, για το τι γίνεται με τις γνωστικές ικανότητες ε, στα παιδιά, καθώς βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τώρα και ψηφιακές τεχνολογίες. Θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην δυνατότητα ο ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός χώρος να είναι κάτι που θα υλοποιηθεί. Εμείς ε, θέλουμε με αναγνώριση των τίτλων σπουδών ε, να υπάρχει ε, περισσότερη ουσιαστικά επικουρικότητα και το θέμα είναι να έχουμε και πραγματική προσθεμένη αξία της Ευρώπης, όχι μόνο τα εθνικά προγράμματα να αναγνωρίζονται. Έχω δύο ερωτήσεις. Είχαμε προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα για την κινητικότητα των φοιτητών και το άλλο η θέση σας για το Discovery U που είναι ε, ουσιαστικά ένα νέο σκέλος του Εράσμους και θέλουμε να το συνδέσουμε περισσότερο με εκπαιδευτικά προγράμματα και να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση που να αφορά μόνο το ταξίδι. Η κυρία Υπουργό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κώστα για τις ερωτήσεις που μου έθεσε. Σίγουρα η πολυγλωσία είναι μια αρχή που την προωθούμε και έχει να κάνει τόσο σε ό,τι αφορά ε, την ε, ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης και ε, μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εθρών. Τώρα, σε σχέση με τις ερωτήσεις σας, συμφωνώ. Πιστεύω ότι οι φοιτητέ μας από όλες τις χώρες θα χαίρονταν πάρα πολύ αν υπήρχε ευρωπαϊκή κάρτα φοιτητών. Γιατί η ελεύθερη κινητικότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία θα διασφαλιζόταν καλύτερα και σίγουρα η δική σας ψήφο στο θέμα αυτό θα μετρήσει πολύ. Από τη δική μου σκοπιά θα το υποστηρίξουμε. Γνωρίζω το πρόγραμμα Discovery U και πιστεύω ότι η προσθήκη εκπαιδευτικών συνιστοσών θα είναι ένα συν στο πρόγραμμα αυτό και θα αυξήσει την ε, αποτελεσματικότητά του. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ για τους ICR. Ε, όχι, δεν θέλετε το λόγο. Η Άλντε. Κύριος Διάκονου. Αν θέλετε. Ευχαριστώ. Εγώ ως κύριος Διακόνου μιλάω, όχι ως μέρος του Άλντε, ως μέρος του φιλελευθέρων. Κύριε Υπουργέ, Πολύ ωραία. Παραθέστε και τον ιστορικό Νικολά Γκιόργκε. Δηλαδή ότι η εκπαίδευση, η παιδεία είναι όσα βλέπεις και όσα ακούς. Και νομίζω ότι είναι σε αυτή η παράθεση, αυτή η πραγματικότητα. Η ερώτηση είναι. Αν μπορείτε να μου πείτε πώς θα βλέπατε να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το πράγμα κυρίως όταν ε, έχουμε τις εξής συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων ε, στον ευρωπαϊκό χώρο. Και αυτό είναι μια άλλη επιθυμία, δηλαδή να είναι συμβατή η διάφορη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική χώροι και φυσικά εφόσον έχουμε μια αγορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται και η παιδεία. Πώς θα το βλέπετε πρακτικά αυτό. Ευχαριστώ κύριε Υπουργός. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Να σα ομολογήσω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τεθεί σε εφαρμογή αυτό που λέει ο Νικόλα Γιώργα, αλλά δεν ε, είναι και αδύνατο να προσπαθήσουμε. Γιατί πιστεύω ότι στην πρωτομάθημη εκπαίδευση, αλλά και όχι μόνο, σε όλους τους εκπαιδευτικού κύκλου, η έμφαση στις θεμελιώδει αξίες ε, με τι οποίε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο ο νέος μαθητής, προκειμένου να διαμορφώσει την προσωπικότητά του, που μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές, να μπορεί να προσαρμοστεί στον κόσμο, και να συνεισφέρει και με τις ε, δικές του δημιουργικές ιδέες είναι μόνο κάποια από τα πράγματα που προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσα στα δικά μας εκπαιδευτικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Χέλγα Τρούπελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να σταθώ στην ε, πολιτική ηγεσία ε, στα πλαίσια της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Άκουσα τους συναδέλφους και όπως είπατε κι εσείς, Υπάρχουν πολλά επιτυχημένα προγράμματα, το Erasmus, το Creative Europe, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους νέους και τους ανθρώπους όπου ζουν στην ύπεθρο σε περιοχές που αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Χρειαζόμαστε τη Ρουμανική Προεδρία να σταθεί υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έτσι ώστε να στηρίξουμε το κοινό μας συμφέρον στην ευρωπαϊκή συνεργασία και στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να συνδράμετε και εσείς και οι συναδελφοί σας στην προσπάθεια αύξησης του προϋπολογισμού προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας για τη συζήτηση αυτή. Και σας διαβεβαιώ, όπως είπα, καταρχήν ως ε, εκπαιδευτικός καθηγήτρια με ενδιαφέρει να υποστηρίξω όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όμως, οι δεσμεύσει ε, που αναλαμβάνει η Ρουμανία κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της είναι πολύ μεγαλύτερες. Επομένως θα υποστηρίξουμε ένα μεγαλύτερο προπολογισμό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπίλτ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί για την ε, επίσημη έναρξη της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ορχήστρα και ουσιαστικά εκτέλεσε τον ύμνο της Χαράς την ένα της Μανία της Ρουμανίας και μια ραψοδία του κυρίου Ενέσκου, του συνθέτη Ενέσκου. Δώσαμε λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα του πλούτου του πολιτισμού μας. Εμείς ε, μοιραζόμαστε μεγάλα έργα και ε, ουσιαστικά τα απολαμβάνουμε ακόμη και αν έχουν παραχθεί από άλλους καλλιτέχνες εκτός της χώρας μας. Λυπάμαι που δεν βρίσκουμε την ίδια ισορροπία στο προγραμματικό έγγραφο της Ρουμανικής Προεδρίας. Αναφέρεται στη σημασία ε, της πρόθεσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης παρουσιάζεται ως ευκαιρία ενίσχυσης τη ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θέλουμε να επιτρέψουμε στον καθένα να μετακινείται παντού στην Ευρώπη για να μάθει, να ανακαλύπτει, να εργάζεται. Όμως τίποτα δεν λέμε για, την, ε, για τον τοπικό πολιτισμό που πεθαίνει. Τίποτα δεν προτείνεται ε, κατά της παγκοσμιοποίησης που τυποποιεί πολιτισμό. Τίποτα δεν λέτε για να έχετε πόλου αριστείας ε, εκτός των μεγάλων Μητροπόλεων. Πολλέ από τι ερωτήσει που ήθελα να σας ε, θέσω ε, έχουν ήδη απαντηθεί γιατί τις έθεσαν οι συνάδελφοι. Όμως για την κινητικότητα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Δεν πιστεύετε ότι πέρα από το δικαίωμα μάθηση και εργασία, οι πολιτεί μα θέλουν να ζουν και στη χώρα του. Να μπορούν να ζουν και στη χώρα του. Σα ευχαριστώ. Κύριε Υπουργό, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπίλντε για την ερώτηση αυτή. Σα σας εξομολογηθώ ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτή την ε, συναυλία, ήμουν στην αίθουσα και την ε, ακόλουθη εβδομάδα έγινε αυτό που είπατε, δηλαδή η κυβέρνηση της Ρουμανίας με κυβερνητική απόφαση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα η οποία, την οποία απολαύσαμε ε, στο Αθήνεο μπορώ να σας πω ότι ίσως ο καθένας ε, με τις δικές τους ε, ρίζες ε, να μπορέσει να συνεισφέρει με τη δική του ενέργεια. Σίγουρα δεν πρέπει να εγκαταλείπτεται το τοπικός πολιτισμός. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις κουλτούρες να αναπτύσσονται. Έτσι λοιπόν ε, δεν έχει πρόθεση η Ρουμανική Προεδρία να παραμελήσει αυτές τις τόσο πολύ σημαντικές στοιχείες για την ανάπτυξη της τοπικής κουλτούρας και την περαιτέρω πρόθεσή τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στον επόμενο Υπουργό, αλλά πριν το κάνουμε έχουμε δύο ακόμα ε, ομιλητές που έχουν στήσει το λόγο. Τζούλου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Υπουργή που βρίσκεται σήμερα εδώ, ε, έχω την Βρετανική επικότητα ε, από την βορειοδυτική Αγγλία και έχουμε πραγματικά έναν ε, τεράστιο πληθυσμό από τη Ρουμανία ο οποίος συμβάλλει στην πολιτισμικότητα της δικής μας περιοχής και θα ήθελα να σας πω ότι όταν έρχονται στη δική μου πόλη, στο Μάντσεστερ και στο Λιβερπούλ, δεν εγκαταλείπουν την εθνική του ταυτότητα. Αντιθέτω, μοιράζονται την ε, πολιτιστική του κληρονομιά και την εθνική του ταυτότητα με εμά. Ε, και έχουμε μία σειρά από ε, εξαιρετικά και πολύ ενδιαφέροντα project και προγράμματα στι πόλει μα, τα οποία ακριβώ συνενώνουν, αν θέλετε, και φέρνουν κοντά ε, όλες αυτές τις διαφορετικές ε, κουλτούρες ε, και όλες τις ιδιαίτερες ταυτότητες, όλες τις διαφορετικές πολιτισμικές εκφράσεις που αποτελούν ακριβώς το μείγμα των διαφορετικών παραδόσεων, των διαφορετικών ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας. Οπότε σας διαβεβαιώ ότι πραγματικά δεν χάνουν την πολιτισμική τους ταυτότητα Ρουμάνοι πολίτες που διαβιώνουν στη δική μας χώρα και αντιθέτως συμβάλλουν στα διάφορα προγράμματα Οπότε από τη δική μου πλευρά αυτό που αναφέρω είναι μια διαβεβαίωση ε, σε ό,τι αφορά τους ερμόνους επόμενους στην Βρετανία και όχι ερώτημα. Παρακαλώ κύριε Υπουργό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Να σας ε, πω ότι όταν βλέπω μια στατιστική ανάλυση στη Ρουμανία, βλέπω ότι πολλοί φοιτητές θέλουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ελεύθεροι να επιλέξουν, όπως είπατε και εσείς. Ε, σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι θα γίνει μετά το Brexit. Όμως ε, μας ενδιαφέρει οι πολίτες ε, να έχουν δικαιώματα που προστατεύονται όπου και να αποφασίσουν να ζουν. Για το Μάτσεστερ και το Λίβερπουλ ήθελα να σας πω ότι ο πρώτος Ρουμάνος που ταξίδευσε με το πρώτο ευρωπαϊκό τρένο Λίβερπουλ-Μάτσεστερ ήταν αυτός που εφήβρε το στυλό πετράκι από ενόρου και στη συνέχεια ήταν κοσμήτερο στο πανεπιστήμιο που σπούδασα εγώ και έγινα και εγώ στη συνέχεια πριν. Σε ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ρόσκο. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση ε, του ε, προγράμματος εργασιών της Ρουμανικής Προεδρίας. Να πω ότι με ευχαριστεί το γεγονός ότι θεωρείτε κι εσείς πολύ σημαντική την πτυχή του περιεχομένου της δασκαλίας. Νομίζω πως ε, θα έχετε ακούσει ε, σχετικά με την σχετική ε, έκθεση που είχαμε συντάξει από κοινού με την κυρία Σοβάσκα σε ό,τι αφορά ακριβώς την ποιότητα της ύλης της διδακτέας. Οπότε νομίζω πως και αυτή η έκθεση μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε περιοχές όπου αυτό δεν συμβαίνει ακόμα. Αξιοποιώντας δηλαδή τις σε πρακτικές. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών ε, ε, προσόντων και διπλωμάτων, εδώ χρειάζονται ακόμα να γίνουν μία σειρά ε, από πράγματα οπότε θα θέλαμε σε σχέση με αυτό να ζητήσουμε την δική σας υποστήριξη. Ε, τρίτον, σε ό,τι αφορά την, τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα της ΕΝΕΣ είναι κάτι που ανέφερε και η κυρία Κώστα και είναι πολύ σημαντικό και σε συνάρτηση με αυτό ε, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές και οι μαθήτρες να διδάσκονται στην μητρική τους γλώσσα. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν και στην ε, δική μου χώρα και πραγματικά θεωρώ πως είναι σημαντικό και στο μέλλον να συνεχίσουμε να προωθούμε την διδασκαλία στη μητρική γλώσσα ε, των παιδιών. Οπότε σας καλώ να υποστηρίξετε και αυτή την πτυχή. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κυρία Υπουργέ, καταληκτικά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Μπόσκορα, Αναμφισβήτητα η συνεχής ε, εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικό ε, στοιχείο για να μπορούν να διδάξουν στην αίθουσα. Και γι' αυτό ε, εγώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχομαι την έκθεση, έχω διβάσει την έκθεση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των διπλωμάτων, η εμπειρία μα δείχνει ότι πολλέ φορέ η άμεση συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων οδηγεί και στην αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων. Νομίζω ότι είναι μία οδό που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε σε ό,τι αφορά την πολυγλωσία. Η Ρουμανία έχει μία εμπειρία βάλτη των πρακτικών. Η Ρουμανία αναγνωρίζει και διασφαλίζει τη διδασκαλία της μητρικής για 20 μειονοτικές γλώσσες και εγώ πιστεύω ότι και νομοθετικά το έχουμε θεσπίσει αυτό και φυσικά θα πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί το να μπορούμε να διαπροστατεύουμε και να διαφυλάσσουμε τη μητρική γλώσσα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Yeah, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Υπουργέ που ήρθατε σήμερα να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας και που απαντήσετε σε ερωτήσεις των μελών. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία για την Προεδρία σας και να επαναλάβω ότι ευχόμαστε να καταφέρετε να πείσετε ε, τους υπουργούς, τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τους υπουργούς οικονομικών, να ε, αυξήσουν την ε, χρηματοδότηση είναι κάτι που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχετε την πλήρη στήριξή μας, ιδιαίτερα για τα προγράμματα τα ε, οποία συζητούμε εδώ στην Επιτροπή και για τα οποία είμαστε αρμόδιοι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ελπίζουμε να καταφέρετε να λύσετε αυτόν τον γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Ταυτότητας, κύριο Βάλερ Ντάνιελ Μπρέας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ. Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών και των δικαιωμάτων δημιουργού που θα επικεντρωθούν στα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με τις κύριες συνιστώσεις του προγράμματος εργασίας μας παρά το γεγονός ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα παράθυρο ευκαιρίας σχετικά περιορισμένο λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών, ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε στις δυνατόν περισσότερους νομοθετικούς φακέλους για να έχουμε αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας αναφέρεται στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τον ε, τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αλλά και τη διασυνοριακή προώθηση των έργων και του ευρωπαϊκού περιεχομένου προτείνουμε να ακουστούν οι φωνές των καλλιτεχνών στην ευρωπαϊκή σκηνή μαζί με την φωνή των πολιτικών και των οικονομολόγων επειδή η δημιουργία και η τέχνη έχουν ε, μία θέση προνομιακή όχι λιγότερο σημαντική από τεχνολογία και το εμπόριο ή δημιουργοί και επαγγελματίε ε, θα πρέπει να μπουν στην καρδιά του ευρωπαϊκού προγράμματος ε, και να μπορούν να αξιολογηθούν οι ευκαιρίες της εποχής του διαδικτύου έχοντας κατά νου τις πιο πρόσφατε ψηφιακές εξελίξεις που άλλαξαν σημαντικά ε, τον τρόπο δημιουργία, διαχείριση και διανομής ε, των πολιτιστικών έργων, η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πεγίωση ανταγωνιστική αγοράς για τους δημιουργούς και του επαγγελματίε του πολιτισμού, αλλά και τη ανάπτυξη νέων μοντέλων επιχειρηματικών ε, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας και θα ελκύσουν μεγαλύτερο κοινό. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δικαιώματα του δημιουργού ε, στο πλαίσιο που ο ε, εξυγχρονισμός του ευρωπαϊκού ε, νομικού πλαισίου αποτελεί κάτι απαραίτητο έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι στον πλούσιο πολιτισμό μας. Η Νουμανική Προεδρία θέλει να υιοθετήσει και την οδηγία δικαιώματος δημιουργού στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Κατά τη ε, διάρκεια των πρώτων εβδομάδων την Ιανουαρίου, η Ρουμανία πρότεινε πραγματικές λύσεις συμβεσμού που περιείχαν τρία στοιχεία. Καταρχήν, την προστασία ε, των συμφερόντων των κατόχων δικαιωμάτων, κάτι που επιτρέπει να λάβουν μια του καλή αμοιβή για τη χρήση των έργων τους ε, σε επιγραμμικά περιβάλλοντα. Δεύτερον, τη διασφάλιση ισότιμα ανταγωνισμού και ευνοϊκών συνδικών ανάπτυξη για τους παρόχου υπηρεσιών και τέλος ε, τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε υψηλό ε, σε υψηλή ποιότητα ε, ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να υπάρχει δημιουργία πλεονεκτημάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες όπως η γνώση του πολιτιστικής ποικιλομορφίας όλων των κρατών μελών και δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές ειδήσει και σε πιο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτή η πρόταση οδηγία είναι όμω ε, ιδιαίτερα πολύπλοκη και τεχνική. Η απόδειξη είναι το γεγονό ότι οι συζητήσει ε, ε, διαρκούν σχεδόν τρία χρόνια. Μπορεί να φέρει πολλά ωφέλη στην νέα ψηφιακή αγορά, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλέ διακλαδώσει. Το Συμβούλιο μα έδειξε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο προβληματισμού για να φτάσει σε μία ενωπημένη θέση. Η Προεδρία θα αναλύσει στη συνέχεια τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον. Μία άλλη προτεραιότητα τη Ρουμανική Προεδρία επίσης ε, αφορά το να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027. Όλοι είμαστε πεπισμένοι για τη σημασία της διασφάλισης της συνέχειας οικονομικής στήριξης για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσει στο να παρέχονται επιχορηγήσει για του καλλιτέχνε και του επαγγελματίε του πολιτισμού. Αν και η πρόοδο στη διαπραγμάτευση του προγράμματο εξαρτάται από τη Συμφωνία για το Πολιτέ Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Προεδρία τη Ρουμανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τι συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τι τομεακέ ενιστώσει ε, των νομοθετικών προτάσεων, χωρί ε, αναφορά στα νούμερα. Θεωρούμε ότι η επίτευξη μια μερική συμφωνία μεταξύ των δύο είναι προς το συμφέρον των κύριων δικαιούχων του προγράμματο μέσω της διασφάλισης μιας εύκολης και προβλέψιμης μετάβασης μεταξύ των δύο γενιών ε, του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τους ε, χρηματοδοτικού μηχανισμούς που είναι βιώσιμοι για το τομεί πολιτισμού και της δημιουργίας, ε, η Ρουμανική Προεδρία θα ενθαρρύνει Επιχειρηματικέ πρωτοβουλίες και μια πιο διευρυμένη χρήση καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότησης. Τα στοιχεία αυτά θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Πολιτισμού που θα λάβει η χώρα στις 16 Απριλίου 2019 στο Βουκουρέστι και θα προσεγγίσει πιθανέ γραμμές δράσης για το μέλλον. Σημαντικά βήματα έγιναν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της εκπόνησης ε, αρκετών μελετών ε, σε σχέση ε, με τα μέτρα χρηματοδότησης ε, των τομέων του πολιτισμού και της βιομηχανία, δείχνοντα τη σημασία ε, καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης όπω είναι οι επιχορηγήσει, τα βάουτσερ, της δημιουργικότητας, τα δάνεια, το κεφάλαιο κινδύνου, τραπεζικές εγγυήσει, το crowdfunding κτλ. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά σε πολιτικό επίπεδο για να δούμε τα μελλοντικά βήματα μια πιθανή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα που να διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διάφορων πηγών χρηματοδότηση, να διευκολύνει την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και να παγιώνει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι ευνοϊκό στην ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και τη δημιουργία. Θέλω επίση να τονίσω το γεγονό ότι η Ρουμανία θα προωθήσει την ε, μουσική και κινηματογραφική ευρωπαϊκή βιομηχανία μέσω τη υιοθέτηση πολιτικών συστάσεων στο Συμβούλιο και τη διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων. Ε, ουσιαστικά η Προεδρία της Ρουμανίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσει μέσω του Music News Europe ε, τη συνεργασία των καλλιτεχνών και την παγίωση ενός ε, ευρωπαϊκού μουσικού ρεπερτορίου. Η διάσκεψη Music Moves Europe θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι στις 21 Ιουνίου 2019 προκειμένου να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ όσων λαμβάνουν αποφάσεις ε, και της μουσικής βιομηχανίας στην Ευρώπη συνεχίζοντας σε μία ε, διάσκεψη για τον ε, τομέα του δικαιώματος του δημιουργού. Σε ό,τι αφορά την γενοματογράφο, θέλουμε να θετήσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου που να αφορούν τη βελτίωση τη διασυνορική κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη συμπαραγωγή. Οι μελέτε δείχνουν ότι γενικά οι, οι συμπαραγωγέ κυκλοφορούν καλύτερα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, γιατί συνήθως ε, διαδίδονται στα κράτη ε, εταίρους. Ε, κάθε έργο δείχνει την επικοινομορφία, την πολιτιστική και την κλωσική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά εκπροσωπεί τα ταλέντα και τις ικανότητες πολλών κρατών μελών και συνεισφέρει στη δημιουργία μιας κοινή ταυτότητα. Οι πολιτικές συστάσεις θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία με των κρατών μελών που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής με τα κράτη ε, όπου έχουμε περιορισμένες ε, γεωγραφικές, ε, περιορισμένη γεωγραφική και χρήση της γλώσσας. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε στις 18-19 Μαρτίου 2019 στο Βουκουρέστι για μια σχετική σύνοδο. Επίσης, Θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε το 2018 με το έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μια κοινή πηγή και θα πρέπει να την ε, συνειδητοποιούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Προεδρία θα τονίσει τη σημασία της προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της διασφάλισης υψηλών προτύπων ποιότητας στην προστασία αυτού και σε παρεμβάσει στον τομέα. Είναι χρήσιμος εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών, αλλά και ε, να ε, μπορέσουμε να παρέμβουμε σε προβληματικές ε, που προκύπτουν όταν έχουμε μείωση της ποιότητας σε περιπτώσεις αποκατάστασης. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε την δημιουργικότητα των νέων γενιών. Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί μέσω της ανάπτυξης δημιουργικότητας ε, της, ε, του καινοτόμου δυναμικού αλλά και της ε, κληροδότησης ε, ικανοτήτων στους νέου προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά έργασία Η Προεδρία θα υπογραμμίσει τη σημασία της νέα γενιά στον πολιτισμό για να αναπτυχθούν ε, διαπολιτισμικέ, δημιουργικέ ικανότητε και ικανότητες επικοινωνίας ε, για την επαγγελματική και προσωπική κατάρτιση προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτε να συμμετέχουν και ενεργά στα κοινά. Αυτέ θα είναι οι κύριε προτεραιότητε τη προεδρία τη Ρουμανία Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσίασή σας. Θα περάσουμε πάλι σε κύκλο ερωτήσεων από τους ε, συντονιστές πρώτα. Κυρία Σόιντροβα, για δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Βέβαια, ο πολιτισμός είναι ιστορική μας ε, και καλλιτεχνική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες, κύριε Υπουργέ. Είναι κάτι που θα πρέπει να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε για τις επόμενες γενιές. Σας ε, καλώ να βρείτε και τους κατάλληλους πόρους για τη δημιουργική Ευρώπη και να επικεντρωθείτε στις προτεραιότητες. Θέλω να αναφέρω την εκπαίδευση στον κινηματογράφο. Γιατί αν μιλάμε για την κινηματογραφική βιομηχανία θέλουμε να έχουμε κοινό, θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που να θέλουν πράγματι να δουν αυτές τις ταινίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε και το σκέλος της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, κάτι που δεν έχει διασφαλιστεί ακόμα. Επίσης, για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, πρέπει να δούμε και το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει διαφοροποίηση, υπάρχουν πολύ περισσότερα προγράμματα στη δύση σχέση, στην ε, δυτική σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Yeah, bitte, Herr Minister κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κυρία Σόντροβα για την ερώτησή σας. Βεβαίως, η πρόσβαση των νέων και συμμετοχή του στην κινηματογραφική βιομηχανία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μια πολύ σημαντική πτωχή στο να εκπαιδευτούν οι νέοι και θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτό να ενέχεται σε μια περίοδο της κατάρτισής τους. Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση, η παιδεία των νέων μέσω του κινηματογράφου, μέσω των όσων παρουσιάζονται στο κινηματογράφο. Τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων θα πρέπει να υποστηριχθεί από πολλές απόψεις. Θα πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση των νέων. Κατά την περίοδο της Προεδρίας, εμείς θα έχουμε κατά νου τις πτυχές αυτές και θα προσπαθήσουμε και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να προσφέρουμε στους νέους ε, μία ως δυνατόν ε, καλύτερη εκπαίδευση και να μπορεί να ε, ουσιαστικά να τους προσφέρει και ένα δημιουργικό σκέλος η εκπαίδευση αυτή. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ε, ευχαριστώ. Μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες οι προτεραιότητε της Ρουμανικής Προεδρίας. Είπατε ήδη πολλά και ξέρω ότι είναι δύσκολε ε, οι τρέχουσε διαπραγματεύσει. Όμω εμεί θα θέλαμε να ολοκληρωθεί σε αυτή τη θητεία. Μιλώ για το copyright. Έχει διαρκέσει τρία χρόνια η συζήτηση, αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Εκτιμώ την πρωτοβουλία της Προεδρίας να κάνει μια απόπειρα να βρει μια κοινή βάση και έχουμε ενθαρρύνει και την ευελιξία εμείς όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με φασιστικότητα, γιατί θα είναι πολύ σοβαρό αν κλείσει αυτή η θητεία, χωρίς να έχουμε νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Γιατί στη συνέχεια θα έχουμε τα κατάλληλα νομοθετήματα, προστατεύουμε και τα δικαιώματα δημιουργού και την πρόσβαση στον πολιτισμό. Τώρα, για το Creative Europe, εγώ είμαι η συγγήτρια. Είπατε κάτι σημαντικό. Στις 20 ε, Φεβρουαρίου εμείς θα γκρίνουμε το κείμενο. Σας ε, επιβεβαιώνω και ελπίζω η Προεδρία να συμφωνεί. Ζητήσαμε αύξηση του προπολογισμού στα 2,8 δισεκατομμύρια γιατί έχει γίνει πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα αλλά δεν έχει αρκετούς πόρους. Μιλήσατε για ενίσχυση και κλείνω για το InvestEU, δηλαδή για διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και θα πρέπει να πλειοπλασιαστούν. Για μας είναι σημαντικό αυτό το θέμα και στο νέο πρόγραμμα InvestEU έχουμε προβλέψει πολύ πιο σημαντικούς δεσμούς, γιατί ουσιαστικά είναι στα μέτρα του κλάδου αυτά τα μέτρα. Επίσης, ε, νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο τον Πολιτισμό και μετά το 2018, που ήταν το πολιτιστικό της κληρονομιάς. Επίσης, εσείς ε, μας ε, μιλήσατε και για το θέμα της συντήρησης και αποκατάστασης. Θέλουμε κοινού κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Υπουργός. Κυρία Κώστα, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας στους τρεις τομείς αυτούς. Καταρχήν, αν μιλήσουμε για την ε, νέα ψηφιακή αγορά, τα δικαιώματα του δημιουργού είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά είναι και ένας πολύ λεπτός φάκελος. Τελευταία είχαμε πάρα πολλές ε, συζητήσεις ε, και παρατηρούμε ότι έχουμε απόκληση απόψεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς είναι τόσο σημαντικό ο φάκελος αυτός, η Ρουμανία θα βάλει τα δυνατά της να τον απεμπλοκάρει το φάκελο αυτό κατά τη διάρκεια τη θητεία αυτής και να δούμε αν είναι δυνατόν μέχρι το τέλος της θητείας να υιοθετήσουμε την οδηγία. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ λεπτό το θέμα. είναι πολύ σημαντικό για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονηθεί ένα κείμενο. Σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργική Ευρώπη, φυσικά είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε για αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Η δημιουργικότητα μπορεί να σημαίνει το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες ειδικές αγορές για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα. σε σχέση με την ε, συντήρηση και αποκατάσταση και την ποιότητα της ε, αναστήλωσης, της αποκατάστασης. Ε, εργαζόμαστε σε διάφορα προγράμματα και θα θέλουμε να έχουμε μία όσο δυνατόν πιο ποιοτική αναστήλωση. Όχι μόνο των μνημείων, δηλαδή να συζητήσουμε τι σημαίνει η αναστήλωση μια πολύ καλή ποιότητα της αναστήλωσης ε, υπάρχει και σε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Είναι κρίμα να μην δίνουμε σημασία στη διαδικασία της αναστήλωσης, είτε μιλάμε για μνημεία, είτε για την αποκατάσταση ενός έργου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Ο κύριος Διακόνου. Ευχαριστώ. Εμείς εργαστήκαμε εδώ πάρα πολύ για ένα θέμα και αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά όλη η Επιτροπή το υιοθέτησε. Το μυαλό μας αφιερώνονταν σε δύο μέρη. Το ένα υλοποιήθηκε το 2018 και το άλλο είναι στα χέρια της ε, Ρουμανικής Προεδρίας, θα έλεγα εγώ, ευτυχώς. Αναφέρομαι στις ε, πολιτιστικές, ε, στρατηγικές, μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να μας αδιαφέρετε κάποια θέματα για την υλοποίηση αυτού του δεύτερου σκέλους. Θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Διακόνο, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Βεβαίως, θα έχουμε κατά νου αυτές τις ε, πτυχές και θα προσπαθήσω να αναφερθώ με κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχήν, όπως είπα και στην παρέμβασή μου, έχουμε την διάσκεψη στη Συγκισοάρα στις 11-13 Απριλίου 2019. Θα προσπαθήσουμε εκεί να εκπονήσουμε κάποια πρότυπα ποιότητα ε, για την προστασία της πολιτιστική κληρονομιάς. Σε σχέση με τη συνέχιση του έτους πολιτιστική κληρονομιάς 2017 και με την ομάδα διαβίβαση ε, των γνώσεων στον τομέα της πολιτικής κληρονομιάς. Οι εμπειρογνώμονε που έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν στη Συγκισοάρα θα ανταλλάξουν βέστιες πρακτικές. Κάτι που είναι απαραίτητο για να υπάρχει μια συνάφεια σε ό,τι αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα της αναστήλωσης και της αυθεντικότητας δεν προσεγγίζονται σωστά. Υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση για να υπάρχουν κάποια κοινά ποιοτικά πρότυπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επανέλθω ε, στο ζήτημα ε, τα δικαιώματα δημιουργού, τα κόπηρα, ε, γιατί είχε συζητηθεί το λόγο ζήτημα πριν από 10 χρόνια και στην ε, διαδικασία μεταρρύθμισης των τελευταίων δυόμιση ετών έχει συζητηθεί ε, επανειλημμένα. Γιατί πρόκειται για, μας, ε, για ένα σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μονοπωλίων και σε ό,τι αφορά το αφήγημα που ακολουθούμε τελικά εδώ, σε ό,τι αφορά τον ορισμό της ελευθερίας. Γιατί αν δεν ορίσουμε με σαφήνεια αυτή την ελευθερία, τότε ισχυρότεροι είναι εκείνοι που επιβάλλονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή μας ε, κουλτούρα ε, και θα πρέπει να καλύψουμε το σχετικό κοινό, όπως ε, προβλέπεται στο άρθρο 13, χωρίς βέβαια να παραβιάζουμε την, τις διάφορες ελευθερίες και την, το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά, και νομίζω πως επαφείτε σε εσά τώρα που αναλαμβάνετε την ηγεσία, υπάρχει το περιθώριο να φτάσουμε σε μια καλή λύση έτσι ώστε να γίνει πιο αποδεκτή η κατάσταση για τους δημιουργούς μας, για τους συγγραφείς μας, για τους ε, εκδότες μας. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχουν ε, πολύ καλές λύσεις επιτάπητος και θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω λοιπόν να κάνετε τις σχετικές διαπραγματεύσεις για να τις ξεκινήσετε από τώρα γιατί εάν αφήσουμε όλα αυτά να τα επιληφθεί το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα προκύπτει. Δηλαδή αυτό που έκανε ο κύριος Βόιτσεκ ήταν ουσιαστικά να φοβήσει τους νέους νέους λέγοντάς τους ότι ε, δεν μπορούν πλέον να κάνουν upload στο YouTube και ούτω καθεξής αλλά δεν είναι αυτή η δική μας προσέγγιση θέλουμε ένα, απλώς και μόνο ένα νομικό σύστημα διοδότησης χωρίς να δημιουργούμε κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ελεύθερη έκφραση και ούτω καθεξής δεν επιβάλλουμε δηλαδή τέτοιου είδους περιορισμού σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το upload την, την αποστολή τη φόρτωση ε, ψηφιακού περιεχομένου. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν αυτά που έχουν αναφερθεί ότι προσπαθούμε δηλαδή να φοβήσουμε τον κόσμο. Προσπαθούμε να βρούμε μια δίκαιη λύση και θεωρώ πως πρόκειται για μια σωστή ρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών και ελπίζω ότι θα συμβάλλετε κι εσείς στην ε, σωστή επίλυση αυτού του θέματος ακολουθώντας ε, ε, τα άρθρα 12 και 13. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Τρούπολ. Άκουσα τα όσα είπατε σε σχέση με τα δικαίωμα δημιουργού. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις, όπως ε, είπατε, ε, μετά από 10 χρόνια, εδώ και 2,5 χρόνια, στι συζητάτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συζητήσεις αυτές μπορούν να συνεχίσουν αιωνίως. Εσείς ε, όμως δώσατε κάποιες διευκρινήσει. Ο δικός μας ρόλος είναι να διατηρήσουμε την ισορροπία θα πρέπει να έχουμε ισορροπίε ό,τι αφορά την προστασία του δικαιώματος δημιουργού αλλά και τη ελευθερία έκφραση. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μία σύγκριση. Όλοι, κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όπως θέλουμε ένας γιατρός να θεραπεύει σωστά έναν αρρωστό, θέλουμε και το ίδιο ένας καθηγητής να παρουσιάζει ξεκάθαρα τις έννοιες. Ε, όταν είναι σε μια θέση το ίδιο πρέπει να κάνει και ο τύπος. Είπαμε προλίγο ότι πρέπει να υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων αλλά και διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Εμείς θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής να κλείσουμε το φάκελο αυτό, διατηρώντας βέβαια μια ισορροπία έτσι ώστε να μπορέσουμε και οι νομοθέτες να ε, έχουμε αυτή την ισορροπία στο νόμο. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα ήθελε κανείς να εδωθεί σαν μια μηχανή λογοκρισίας. Η ισορροπία λοιπόν είναι πολύ σημαντική και ο δικός μας ρόλος διαμεσολαβητή είναι ακριβώς να διασφαλίσει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Julie Ward. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σημείωσα ότι στην αρχή της ομιλίας σας είπατε πόσο σημαντικό είναι να ακούγονται οι φωνές των καλλιτεχνών. στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ ίδια είμαι καλλιτέχνητα, μάλιστα πρωτού γίνω πολιτικός και Συμμερίζομαι λοιπόν τον Ντέμιαν Τρεχίχη. Έχουμε και δύο αυτήν την διπλή ταυτότητα, ο οποίο είναι μέλο της ε, επιτροπή Πολιτισμού. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ενεργοί και προσπαθούμε να καταστεί δυνατό να ακούγεται η φωνή του καλλιτέχνη εδώ, ιδιαίτερα ε, των νέων καλλιτεχνών, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να βιοποριστούν από την τέχνη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και η Χέλκα για την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού. Και να αναφερθώ στις ε, ευκαιρίες που υπάρχουν. Μία από αυτές είναι ότι η κοινή ε, συνελεύση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα γίνει την Ρουμανία, στο ε, Σινάι, μαζί με ένα συνέδριο για την ε, νεολαία. Και θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο και να δώσουμε ε, όθηση στον διαπολιτισμικό διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Ακουόρτ. Εκτιμώ τα όσα είπατε εδώ. Μιλώντας για τους καλλιτέχνες είπατε ότι προέρχεστε από αυτόν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Εγώ βλέπω ε, ότι για να είναι κάποιος ένας καλός καλλιτέχνης ε, πρέπει να έχει ταλέντο. Και λένε ότι με το ταλέντο γεννιέσαι, δεν μπορείς να το αποκτήσεις ε, μέσω της εκπαίδευσης. Πρέπει να κάνουμε να ακουστούν οι φωνές των καλλιτεχνών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα κάθε καλλιτέχνης ε, να μπορεί να παρουσιάζει το έργο του και να τον υποστηρίζουμε και να τον προστατεύουμε. Η προστασία των καλλιτεχνών και του δικαιώματος δημιουργού είναι ένα θέμα που θα είναι προτεραιότητά μας στην περίοδο αυτή. Στη Σινάια θα λάβει χώρα με πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι πολύ καλή η πρότασή σας και θα τη λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο σε αυτόν τον κύκλο ερωταπαντήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Υπουργό που μα παρουσίασε το πρόγραμμα τη Προεδρία και απάντησε σε όλε τι ερωτήσει. Σα ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην ε, Προεδρία σα και πέρα από αυτή. Περνάμε τώρα στον ε, τελευταίο ε, προσκεκλημένο Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού Κόνσταντιν Μπόγκταν Ματέη. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, εξέτοιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Είναι τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας για τον τομέα του αθλητισμού και της νεολαίας. Στο τομέα της ε, νεολαίας η πρώτη προτεραιότητα που έχουμε ε, έχει τίτλο «Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες για τους νέους». Ε, κατά το όραμα της Ρουμανικής Προεδρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο ευκαιριών όπου θα έχουν πρόσβαση ισότιμα όλοι οι νέοι χωρίς καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων εντάσσονται πιο σημαντική που θα διαχειριστεί η Ρουμανική Προεδρία στον τομέα της νεολαίας. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Εράσμους. Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφιερώνεται στη νεολαία. Έχοντας ε, κατά νου το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έκλεισαν με επιτυχία πέρσι, και έχοντας κατά νου τα λίγα στοιχεία καινοτομία ε, των νέων προτάσεων, μπορούμε να πούμε ότι δεν ε, θα έπρεπε να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δύο συνομοθετών. Θεωρούμε επίσης ότι σε ένα επικοδομητικό κλίμα και σε ένα ρεαλιστικό κλίμα μπορούν να γίνουν, μπορεί να γίνει σημαντική πρόοδος σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις επί όλων των μη δημοσιονομικών πτυχών ε, των προτάσεων του προγράμματος πλαίσιο αυτό το θετικό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ρουμανική Προεδρία είναι έτοιμη να προχωρήσει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο δυνατόν ε, περισσότερο σε αυτούς τους σημαντικούς φακέλους. Πάμε τώρα στο μη νομοθετικό σκέλος ε, σε ό,τι αφορά τη θητεία της Ρουμανικής Προεδρίας. Θα ξεκινήσει η εφαρμογή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ένα νέο διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους νέους που αντικαθιστά το διαθρωμένο διάλογο ένα τίτλο που ίσχυε μέχρι πέρσι. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε μαζί με τον ευρωπαϊκό τομέα της νεολαία ε, να προωθήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με του νέου και να συνεισφέρουμε στην αύξηση του βαθμού εκπροσώπηση στη διαδικασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των νέων της Ευρώπης ε, από όλε ε, τις ε, κοινωνικονομικές κατηγορίες θα ακουστεί. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω το πρόγραμμα εκπρόσωπος νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί η ενεργή συμμετοχή δύο εκπροσώπων των νέων της Ρουμανίας στις δραστηριότητες πρόθεσης και άσκησης της Ρουμανικής Προεδρίας στον τομέα της νεολαίας. Επίσης, η Ρουμανική Προεδρία θέλει να συνεισφέρει στην ε, αύξηση της ποιότητας του διαλόγου μεταξύ των δημοσίων αρχών και των νέων, καθώς ε, και στο να φέρει τους νέους πιο κοντά στο ε, έργο, στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαβουλεύσεις ε, με τους νέους που έχουν ε, υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις Βρυξέλλες μας έχουν ε, δείξει ότι η ένταξη στην αγορά εργασία είναι μία από τι κύριε ανησυχίε των νέων σε σχέση με το μέλλον του. Μπορούμε να περιμένουμε πιο συγκεκριμένα ότι σε 15-20 χρόνια θα έχει διαφορετική μορφή εργασία. Με την έννοια ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα των δημογραφικών εξελίξεων, τη κλιματική αλλαγή ή της τεχνολογικής πρόοδου. Ενώ η σημερινή δυναμική της αγοράς εργασίας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για την ε, απόκτηση της πρώτης θέσης εργασίας από τους νέους. Πολλοί εξ αυτών ε, κινδυνεύουν να μείνουν μπλοκαρισμένοι μέσω πρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα σε προσωρινές θέσεις εργασίας ε, με περιορισμένη κοινωνική προστασία και με περιορισμένες ευκαιρίες ε, να ε, έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και βλέπουμε να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και ένα φαινόμενο που αποκαλείται στα αγγλικά in work poverty. Η δραστηριότητα των ναι, νέων, η άτυπη εκπαίδευση ή ο θελοντισμός ε, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ε, ουσιαστικά τομείς όπου θα αναπτύξουμε πολιτικές και παρεμβάσεις που να διασφαλίζουν μια επιτυχή μετάβαση των νέων προς αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σήμερα και αύριο. Έτσι λοιπόν το κύριο θέμα που προτείνει η Ρουμανική Προεδρία στον τομέα της νεολαίας αναφέρεται στην αύξηση της προσαρμοστικότητα των νέων για την αντιμετώπιση ε, των ε, μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα εργασία. Θα προτείνουμε λοιπόν ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά επιπρόσθετα όταν μιλάμε για το μέλλον της εργασίας. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε προοπτικές, ιδέες και λύσεις από την πλευρά των νέων, γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή των τεράστιων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην ε, αγορά εργασίας. Η διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νεολαία, ένα ε, σημαντικό γεγονός ε, στο πλαίσιο του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο που θα οργανωθεί στο Βουκουρέστι στις 25 έως τι 28 Μαρτίου θα προτείνει στους νέους ε, αυτό το θέμα προβληματισμού προκειμένου να τους προκαλέσει να παρουσιάσουν οι ίδιοι και λύσεις για αυτή την ανησυχία που είναι και δική τους και δική μας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Τώρα, να μετακινηθούμε στον τομέα του αθλητισμού. Ένα από του στόχου κλειδί της Ρουμανική Προεδρίας είναι η παγίωση μια Ευρώπη κοινών αξιών. Μεταξύ αυτών των κοινών αξιών αισθανόμαστε ε, ότι είμαστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με την πρόθεση της αλληλεγγύης και της ισότητας ε, των ευκαιριών. Έτσι, η πρώτη προτεραιότητα που προτείνει η Προεδρία της Ρουμανίας αναφέρεται στην πρόσβαση στον αθλητισμό για τα άτομα με μειωμένες ευκαιρίες. Δεν θα αναφέρω το προηγούμενο μήνυμα ε, σε σχέση με το πρόγραμμα Εράσμους, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, διάσταση της ε, κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Και για το λόγο αυτό βρίσκεται και ένα τμήμα του Εράσμου σε αυτές τις προτεραιότητε. Ένα θέμα που θέλουμε επίσης να διερευνήσουμε στι δραστηριότητέ μα στον τομέα του αθλητισμού αναφέρεται στη διευκόλυνση της πρόσβαση στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίε. όπου σκοπεύουμε να εθετήσουμε ένα σύνολο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρακτικά προτείνουμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που εμποδίζουν ε, τη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών σε αθλητές εκδηλώσεις και θέλουμε να προωθήσουμε μέτρα που να μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ζωής ε, των ατόμων με αναπηρίες ε, σε στο μέσο του αθλητισμού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων σκοπεύουμε να οργανώσουμε στις 14 Ιουνίου στην Κωνσταντσα μια διάσκεψη για τον αθλητισμό και τα άτομα με μειωμένες ευκαιρίες και φυσικά εκεί θα συζητηθεί και το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Στο σημερινό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά το πρόβλημα του ντόπινγκ, της φαρμακοδιέργησης ε, και ε, των ε, ελλείψεων ε, που βλέπουμε στους κανονισμούς αντιτόπικ όπου εμπλέκονται αθλητές και ακόμη και ομοσ... αθλητικές ομοσπονδίες αλλά και εθνικοί φορείς είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνουμε σημαντικέ προσπάθειε για να καταπολεμήσουμε τη φαρμακοδιέργεση. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν ε, αυτέ τι συζητήσει, συνεισφέροντα με μια ισχυρή φωνή ε, στι ε, συνεδριάσει του Παγκοσμίου Οργανισμού κατά τη φαρμακοδιέγερση. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιτυχία επιτυχία της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Ξεκινούμε τώρα με τον ε, νέο γύρο Ρωτήσω και απαντήσω, Οπότε δίνω πρώτο λόγο στην κυρία Σόντροβα για δύο λεπτά κατά το μέγιστο. Ναι. Υπάρχει, ε, όπω γνωρίζετε, μια νέα νομοθεσία, ο νέο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη ε, που συζητείται. Πρόκειται δηλαδή για μια ε, νομοθετική διαδικασία. Ελπίζουμε πω θα έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επίπεδο διαπραγμάτευση δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έω το Μάρτιο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα εδώ να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δικής σας ε, προεδρίας. Ε, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία αυτού του προγράμματος ε, και, την, και τον σχετικό πληθυσμό των 30 ετών, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετάχουν στις δράσεις αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Σότροβα και σας διαβεβαιώ ότι θα έχετε πάση υποστήριξη από εμάς. Χαίρομαι που έχουμε τις ίδιες ε, ιδέες ε, και όταν μιλάμε και για την ηλικία, τα 30 έτη. Σας διαβεβαιώ ότι θα σας υποστηρίξουμε πλήρως και είμαι επιβεβαισμένος ότι θα καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες από κοινού για να πετύχουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εκτίμησα το γεγονό ότι εσεί ε, θέλετε να έχετε μια εγκάρσια προσέγγιση για τι ίσε ευκαιρίε ε, και την ένταξη σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για του νέου, δηλαδή όχι μόνο στα ειδικά προγράμματα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση. Και εμεί είμαστε πολύ προσεκτικοί για τη διάσκεψη των νέων ε, και Πάντοτε ε, θέλαμε να προωθήσουμε ένα νέο διάλογο με τους ε, νέους. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε καλύτερα πώς. Τώρα, για το σώμα αλληλεγγύης. Ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια. Εμάς μας ενδιαφέρουν τρεις διαστάσεις. Καταρχήν, πάντοτε να υπάρχει μια διεθνική διάσταση σε σχέση με το τι κάνουν τα παιδιά ακόμη και μέσα στη χώρα τους. Το θέμα της ε, πρόσβασης είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους που προέρχονται από ένα μεταναστευτικό background και το τρίτο είναι ε, το θέμα των ε, καθηκόντων και της ευθύνης που έχουν αυτές οι οργανώσεις που οργανώνουν τα προγράμματα Ουσιαστικά θέλουμε να στρέφεται κυρίως στον αθελοντισμό και στην ενεργή συμμετοχή του πολίτη το πρόγραμμα αυτό, αλλά θα θέλαμε και ένα σκέλος κατάρτιση στην εργασία. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία ουσιαστικά οικοδομεί την ε, ιδιότητα του πολίτη από τα κάτω. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος με τους νέους. Θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερες συζητήσεις και συναντήσεις με τους νέους και βεβαίως από κοινού να βρούμε λύσεις για την επιλύση των προβλημάτων. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τις λύσεις με τις οποίες θα έρθουν αυτοί προς τα μας, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και εμείς θα πρέπει να έρθουμε να τους συναντήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με όσα είπατε και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα διάλογο μας δυνατόν περισσότερους νέους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Διάκονου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που θέλετε να συνομιλήσετε με τις νέους. Λυπάμαι, εγώ δεν είμαι νέος. Ας κάνετε ένα διάλογο και με έναν ηλικιωμένο. Δεν υπάρχει δυστυχώ ε, Υπουργείο Τρίτη Ηλικία όπω υπάρχει για την νεολαία, αλλά τέλο πάντων τα καταφέρνουμε. Στην αρχαία Ελλάδα, ε, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών ε, Αγώνων, σταματούσαν οι πόλεμοι μεταξύ τους προκειμένου να προβούν σε αθλητικές δραστηριότητες. Τίποτα δεν έχουμε μάθει από αυτό. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε δυστυχώς ε, διάφορους πολέμους και συγκρούσεις που τους βλέπουμε ακόμη και στα στάδια. Έχαμε στην διάταξη και ένα παρόμοιο θέμα που ξεκινά από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εμείς δίνουμε μόνο συμβουλευτική γνωμοδότηση. Σας προτείνω λοιπόν ε, η Ρουμανική Προεδρία να δώσει προσοχή και στο θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θέμα της ασφάλειας ε, στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και κυρίως στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Είναι ένα καυτό θέμα και μας ενδιαφέρει όλους. Σας ευχαριστώ. Έτσι, Νέους και γέρους. Ja, vielen herzlichen Dank. Ευχαριστούμε. Ε, αν οι οικογένειε δεν μπορούν πλέον να πηγαίνουν στο γήπεδο, βέβαια όλοι μα θα έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ. Ναι, βέβαια είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί. Με ανησυχεί και γιατί εγώ ουσιαστικά έχω σπουδάσει ε, γυμναστής και γνωρίζω και τα προβλήματα ε, στα διάφορα στάδια. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες ε, για να προληφθούν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή να υπάρχει σωστή επίβλεψη των ε, σταδίων ε, μέσω καμερών παρακολούθησης και υποδομής. Είμαι εμπισμένος ότι θα καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες για να μπορέσουμε να προλάβουμε ε, τέτοια φαινόμενα. Εμείς ανησυχούμε στη Ρωμανία για τέτοια φαινόμενα όπως γνωρίζετε στη Ρουμανία θα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2020. Έχουμε σχετική εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι για να οργανώσουμε μια τέτοια ε, πολύ σημαντική εκδήλωση και είμαι σίγουρος ότι θα διασφαλίσουμε και ένα καλό κλίμα για όσους θέλουν να έρθουν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ε, και αναφέρομαι στο γύρο 2020. Και σας ε, στέλνω από τώρα την πρόσκληση να είστε κι εσείς ε, εκεί στο στάδιο και να παρακολουθήσετε τους αγώνες για το Euro 2020. Σας ευχαριστώ. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Αξιότιμη κύριε Υπουργή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια προσωπική ε, εμπειρία. Είχα εργαστεί από κοινού με τον Ευόγνε στην Επιτροπή Αγκρή και ε, θα ήθελα να διαβάσετε στη συνάδελφο τα ε, χαιρετίσματά μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική σας προεδρία, να πω ότι έχετε να παίξετε ένα ε, πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, δηλαδή εκείνο που καλείστε ε, να κάνετε είναι να προσπαθήσετε βέβαια να μειώσετε το χάσμα ανάμεσα και στους φτωχότερους και τους πλουσίους καθώς βλέπουμε αυτήν την τάση να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, ε, είδαμε ότι υπήρχε μια αναφορά ε, σε ό,τι αφορά τα New Skills στην ε, ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο θεματολόγιο τη και βλέπουμε ότι η δική σα Προεδρία ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την εξέβρεση θέσεων εργασία για του νέου. Πράγμα το οποίο αφορά και μια πρόσφατη γνωμοδότηση που συνέταξα. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιε είναι ακριβώ οι πρωτοβουλίε που θέλετε να αναλάβετε έτσι οι νέοι να μπορούν να κάνουν επιτυχώ τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά αγορά εργασία. Θα χρειαστεί προφανώ να γίνει επένδυση των καταλήλων ε, πόρων ε, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αλλά θα ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά ε, το πώ ακριβώ σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα σχετικά κονδύλια και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus για αυτήν τον τομέα. Επίση, κάτι ακόμα, πώ θεωρείτε πώ θα μπορούσε να διαρθρωθεί ένα διαρθρωμένο διάλογο με του νέου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω. μας ανησυχεί πολύ το τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χαιρόμαστε που ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού θα δοθεί για την εξάλληψη κάποιων προβλημάτων και για την καταπολέμηση της ενεργείας. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους νέους ε, για να περιορίσουμε στο δυνατόν την ανεργία των νέων. Όμως, όπως ε, είπαμε, για όλα αυτά χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη δική μας ε, συμμετοχή, να έχουμε συνεχή κονδύλια που θα το διοχετεύουμε σε αυτόν τον τομέα έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ενεργεία των νέων. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι από κοινού θα καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε χαμηλότερη ενεργία στους νέους. Και Επίσης, ε, μια πολύ σημαντική πτυχή έχει να κάνει με τις ψηφιακές δεξιότητες ε, που θα πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι και θα πρέπει και εμείς να εργαστούμε σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ward, Ευχαριστώ πολύ. Julie Ward, ένα λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ πως οι νέοι είναι το κλειδί που θα αποφασίσει αν εμείς ε, θα δημιουργήσουμε ένα επιτυχημένο οικοδόμημα ή όχι. Η ενέργειά τους και οι φρέσκες ιδέες τους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όμως ε, οι νέοι δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με μας και δεν αναφέρομαι στους ε, νόμους αλλά στις πολιτισμικές νόρμες. Ορισμένες φορές έχουμε μία εικόνα του πολιτισμού πολύ στενή. Όμως υπάρχουν πολλές ε, νέες υβριδικές μορφές ε, του πολιτισμού και της τέχνης. Υπάρχει η τέχνη του δρόμου, η, ε, το παρκούρ που είναι έτσι μια διασταύρωση αθλητισμού και τέχνης αν θέλετε και νομίζω πως πρέπει να είμαστε περισσότερο προ ορατική και πιο ανοιχτόμυαλη στις τέχνες και τους νέους και τον πολιτισμό και να μην αποκλείουμε μορφές τέχνης και μορφές πολιτισμού που είναι έξω από το συνηθισμένο. Να δίνουμε την κατάλληλη προσοχή και την κατάλληλη οικονομική στήριξη ε, στους νέους για την τέχνη που εκείνοι θέλουν να δημιουργήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Βεβαίω, συμφωνώ μαζί σα ε, ότι ο πολιτισμό και η τέχνη παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην κατάρτιση των νέων. Και ακριβώ ε, επειδή είμαι και υπουργό νεολαία και αθλητισμού και ο αθλητισμό έχει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων και νομίζω ότι και αυτά τα τρία μπορούν να τεθούν στην ίδια κατεύθυνση για να μπορούμε να συνεισφέρουμε. Επίση, είμαι επιπισμένο ότι μαζί με του συναδέλφου, ε, την Υπουργό Παιδεία και τον Υπουργό Πολιτισμού, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τους τρεις αυτούς κλάδους και να διοχετεύσουμε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να ευχαριστήσω ξανά και τους τρεις υπουργού που ήρθαν σήμερα στην Επιτροπή μας και κλείνοντας θα ήθελα να πω δύο λόγια για ε, το Γενικό θέμα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, για τους ε, φακέλους ε, για τους οποίους είμαστε αρμόδιοι και συνδεδεμένοι η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 ε, με τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και Ήτρε. Η... πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα μέρος του στόχου έστω με το Συμβούλιο έτσι ώστε να καταφέρουμε σε πρώτη ανάγνωση να εγκρίνουμε ένα κομμάτι του πακέτου. Ε, νομίζω πως χωρίς να ανακαταψουμε και άλλε επιτροπέ, θα πρέπει τουλάχιστον εμείς εκεί που είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ε, πέρα όμω από τι πρακτικές δυσκολίες και την τεράστια πίεση χρόνου που υπάρχει, υπάρχουν ε, και θέματα στρατηγικής ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ο χρυσός κανόνας είναι ο εξή τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να επιτευθεί η συμφωνία. Και πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, αλλά να μην είμαστε βιαστικοί, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να δούμε τι ε, χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα και για ποια προγράμματα. Ε, χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή ε, Χρειαζόμαστε σε ορισμένα προγράμματα πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την υφιστάμενη. Ε, σε ορισμένα προγράμματα πρέπει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση μάλιστα. μάλιστα. Και μάλιστα στην περίπτωση του Εράσμους οφείλουμε να συζητήσουμε και με την Ρουμανική Προεδρία και θα ήθελα να το κάνουμε αυτό. Τώρα, Επίσημε ή ανεπίσημε διαπραγματεύσει δεν έχουν καμία σημασία αν τα αποτελέσματα είναι ελλειπή. Σε ό,τι αφορά το Εράσμου και το Δημιουργική Ευρώπη, το ζητούμενο είναι αν θα λάβουν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. Ε, αποφασιστικό είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών και σε ό,τι αφορά το Εράσμου, ε, νομίζω πω πρέπει να συζητήσουμε και τα νέα προγράμματα που έχουν προταθεί στο πλαίσιο αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε όμως πρώτα για τη χρηματοδότηση πριν μιλήσουμε για το περιεχόμενο. Αν δεν ξέρουμε τι χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Να καταστεί σαφέ αυτό. Το συζήτησα και με τους υπουργούς και με ε, τους ε, πρέσβεις αυτή την τελευταία εβδομάδα. Δεν ε, βέβαια θέλω να δείξω δυσπιστία προς την Ρουμανική Προεδρία, αλλά βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατάθεση την πρότασή της σχετικά αργά και τώρα εμείς πρέπει να δούμε αν μπορούμε, αν προλαβαίνουμε μάλλον στο Κοινοβουλίο να ψηφίσουμε το φάκελο αυτό σε πρώτη ανάγνωση έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα χρόνου. Όμως η Ρουμανική Προεδρία θα είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά, που θα ε, καταφέρει ή όχι να λύσει το χώριο δεσμό και να ξεμπλοκάρει το θέμα της χρηματοδότησης. Μόνο τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε ε, επί του περιεχομένου. Και ελπίζω να το καταφέρουμε, να το καταφέρετε εσείς ε, καλύτερα από τις προβλέψεις. Θα ήθελα λοιπόν να το πω αυτό έτσι ώστε να μην δημιουργείται η εντύπωση πω εμεί δεν θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε πριν γνωρίζουμε πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά που ήρθατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία ε, για την Προεδρία σας, η οποία έχει έρθει σε μια δύσκολη στιγμή. Σα εύχομαι λοιπόν ξανά καλή επιτυχία για του ερχόμενου έξι μήνε και καλό μεσημέρι.